<clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Χαίρετε, ιδίως σε όσους μόλις ήρθαν, με χαρά υποδέχομαι έναν συνήθι παρόντα στη συνεδριά μας, τον κύριο Αλέξανδρο Ρόντο, ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κέρα της Αφρικής. Δεν ξέρω αν είναι δυστυχώ ή ευτυχώ που το κέρα τη Αφρική αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα λόγω των γεγονότων στο Σαχέλ και το Μαλί. Παρ' όλα αυτά, η περιοχή αυτή από πολλές απόψεις έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δράση της Ένωσης, τη δράση που επιχειρεί συλλογικά να φέρει σε πέρας αυτήν την ε, περίφημη σφαιρική προσέγγιση. Θα ξέρεις αλλά δεν υπάρχει ούτε μία ομιλία της υπάτης εκπροσώπου που να μην υμνεί την ε, σφαιρική προσέγγιση στη δράση της Ένωσης στην Αφρική. Τώρα βέβαια να δούμε σε τι βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα την οποία ζει επιτόπου ο ειδικό εκπρόσωπος θεσμικά και ε, από πλευράς κάθε διάστασης της δράσης μας. Σίγουρα υπάρχει ε, μεγάλη συγκέντρωση μέσων προσωπικού αλλά και αποστολών στρατιωτικών και πολιτικών σε αυτό το τμήμα της Αφρικής και να δούμε βέβαια αν θα το επιβεβαιώσετε αλλά θεωρούμε ότι όλα αυτά έχουν κατορθώσει να επιτύχουμε μια σχετική επιτυχία και θα ξέρετε ότι ο πρόσφατα εκλεγμένος ε, πρόεδρος της Ομαλίας ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και ε, μας μίλησε για μια σχετική εξομάλυνση. Εμένω σχετική γιατί αν θυμηθούμε το παρελθόν της Σομαλίας ε, δύσκολα θα μιλήσουμε για ομαλή κατάσταση αλλά έχει υπάρξει πρόοδο σε θεσμικό, οικονομικό, στρατιωτικό επίπεδο. Αυτές οι πρόοδοι πρέπει βεβαίως να εδρεωθούν και με χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις σας. Εποφελούμε προσθέτοντας πω ότι πριν από μερικέ μέρες ψηφίστηκε ένα ψήφισμα που επιμικίνει την ε, θητεία και εντολή τη ΜΙΣΕΜ, της Αφρικανικής Δυναμή. Έγινε πολλή συζήτηση γι' αυτό, αν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει από την παρούσα σύσταση, αν θα πρέπει να γίνει ειρηνευτική αποστολή των ΗΕ. Ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί προκύπτει και για μια άλλη περιοχή, το Μαλί. Ποια διδάγματα μπορούμε λοιπόν να εξαγάγουμε από την ε, πείρα μας στη Σομαλία για άλλες περιοχές της Αφρικής. Και αυτό ενδιαφέρον θέμα συζήτησης. Και υπάρχουν ε, πολιτικά, διπλωματικά γεγονότα που ε, θα λάβουν χώρα για τη Σομαλία τον ε, Μάιο θα γίνει μια διάσκεψη στο Λονδίνο και προβλέπεται και μια διάσκεψη εδώ τον Σεπτέμβριο όπου θα υπάρξει πολλή εκπροσώπηση για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σταθεροποίησης της χώρας. Η Σομαλία είναι βέβαια η προτεραιότητα της εντολής σας, αλλά στο κέρας της Αφρικής ε, είδαμε και εκλογικά γεγονότα στην Κένια πρόσφατα. Ίσως και εδώ να μπορείτε να μας πείτε τι επίδραση μπορεί να έχει στις πολυμερείς προσπάθειες που γίνονται για τη Σομαλία. Και Φυσικά υπάρχουν και τα θέματα του Σουδάν ε, επί του οποίου για ευνόητους λόγους ε, δεν αναλαμβάνεται πολλές ε, δραστηριότητες αλλά και το θέμα του Νείλου, οι σχέσεις Αιθιοπίας-Αιγύπτου επ' αυτού, θέμα ζωτικής στρατηγικής σημασίας που μας το κρύβουν οι συγκρούσεις. Αλλά το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι διαρθρωτική σημασία για την περιοχή. Δίχως άλλα, Αλέξανδρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αγνώ. Με χαρά επανέρχομαι ενώπιόν σας. Ας προσπαθήσω να αναφερθώ σε διάφορα θέματα, ορισμένα τα ανέφερε ο Αγνώ ήδη. Πρώτα απ' όλα, ας ε, δούμε το πρόσφατο παρελθόν. Διορίστηκα πριν από λίγο πάνω από ένα χρόνο. Άρα έχω την ευκαιρία πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη που όλοι μου δίσατε, μου δώσατε συγγνώμη. Συζήτησα με πολλούς είτε σε συναντήσεις είτε μεμονωμένα, ανταλλάξαμε απόψεις και με, βοήθησα, με βοήθησε πολύ η πείρα που απεκόμισα. Η... Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νομοθετικές αρμοδιότητες και μπορεί να δημιουργήσει ουσιώδη πολιτική, ουσιώδη μέσα στήριξης της Ένωσης. Δύο-τρεις εισαγωγικέ παρατηρήσεις για την περιοχή. Πρώτον, Σκεφτείτε το κέρα της Αφρικής. Ένα σύνορο ο Νείλος, το άλλο σύνορο Ερυθρά θάλασσα, Δυτικός Συνδικός. Αυτά είναι τα δύο θεμελιώδη σύνορα που εμπεριέχουν το κέρα της Αφρικής. Υπάρχουν ε, βεβαίως σχέσεις και εμπόριο και πέραν των σύνορων αυτών, αλλά σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να συγκεντρώσετε την προσοχή σας. Στην περιοχή αυτή έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες μεταβάσεις, αλλαγές τον τελευταίο χρόνο. Η Σομαλία συμπλήρωσε την τυπική μετατροπή της, αλλά τώρα είναι σε φάση ουσιώδους μετατροπής σε κανονικό κράτος. Είναι σε πρώτη φάση βέβαια. Ναι, μένει είμαι αρκετά θετικός, αλλά είναι σχετικό αυτό. Αλλά είμαι θετικός. Και χαίρομαι που μπορέσατε να ακούσετε τον πρόεδρο που προσπαθεί η χώρα του να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Κένια μόλις έκανε εκλογέ. Αν εξετάσετε όλες τις επιλογές που υπήρχαν, ο τρόπος που έγιναν ε, οι εκλογές τελικά ήταν από τις ε, καλύτερες λύσεις. Ήμουν παρόν και συγκινήθηκα όταν είδα ένα έθνος να προσφεύγει ειρηνικά, ήσυχα, περιμένοντας για ώρες μπροστά στα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν. Πολλοί δικοί μας πολίτες ε, μπορεί και να είχαν φύγει, αλλά εκείνοι περίμεναν. Αυτό λοιπόν με εντυπωσίασε. Και η Αιθιοπία είναι σε φάση μεγάλων αλλαγών. Πέθανε ο Μέλες, που ήταν ε, διανοητικά κορυφή στην περιοχή και η επιρροή του ξεπερνούσε κατά πολύ τα σύνορα της χώρας του. Και εδώ υπήρξε μια σταδιακή μετάβαση. Τι θα προκύψει, περιμένουμε. Αλλά έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι η αλλαγή αυτή γίνεται ειρηνικά. Στα κράτη στο Σουδάν τουλάχιστον δύο χώρες προσπαθούν να βρουν τρόπο να συμφωνήσουν. Σε τι να συμφωνήσουν. Η καθεμία έχοντας σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά ακόμη πρέπει να γίνει μεγάλη πρόοδος. Και δεν αναφέρομαι καν στο πώς διοικούν τη χώρα τους. Το ζήτημα είναι πώς διεξάγουν τις σχέσεις τους ακόμη. Αλλά επειδή σε αυτή την περιοχή που όλοι θεωρούμε ότι είναι πηγή βαθιών αιτιών αστάθειας. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή και έχω και την πύρα των Βαλκανίων ε, στο μυαλό μου που μεταφέρω. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή κάποια στιγμή καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι το να θυσιάσουν ένα τμήμα από τα συμφέροντά τους για το κοινό καλό είναι πιο θετικό από την ε, σκληροτράχυλη επιδίωξη του στενά εννοουμένος, ε, στενός εννοουμένος καλού του. Για πρώτη φορά οι Υπουργοί Εξωτερικών είπαν ότι πρέπει οι χώρες να επιλύσουν τις διμερείς συγκρούσεις τους και να υπάρξει περισσότερη περιφερειακή ενοποίηση. Έτσι λοιπόν έχω περισσότερα επιχειρήματα για να συζητήσω μαζί τους. Αλλά παρόμοια ήταν τα πορίσματα και της ε, συνάντησης κορυφής της, ε, του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας. Και πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να το συζητάμε με την Αφρικανική Ένωση. Αλλά υπάρχει μια αλλαγή αντιμετώπισης, ότι το κόστος δηλαδή της έλλειψης ενοποίησης, της έλλειψης συνεργασίας δεν αξίζει πια να φέρετε. Ας ε, περάσω τώρα πιο αναλυτικά σε ορισμένα σημεία της περιοχής. Στη Σομαλία από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη έχουμε την απαρχή της διαπίστωσης των καρπών μιας πολιτικής που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη ασφάλεια σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα της χώρας. Όχι βέβαια παντού. Η Al-Shabaab εξακολουθεί να ε, λειτουργεί σε ορισμένα τμήματα της χώρας, αλλά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια στρατηγική ασφάλειας που επέτρεψε να υπάρξει και πολιτική. Και οι Σομαλοί έχουν ε, σε αυτή τη φάση την αίσθηση ότι εκπροσωπούνται περισσότερο στην πρωτεύουσά τους από ότι ε, οποτεδήποτε στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι απομονωμένες περιοχές της χώρας που ζούσαν σε αυτάρκεια σταδιακά επανέρχονται σε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο. Γίνονται λοιπόν ε, πολλαπλές τοπικού επίπεδου διαπραγματεύσεις και πρέπει να τις ενθαρρύνουμε γιατί οι Σομαλοί βέβαια ξέρουν πώς να συνομιλήσουν ένας με τον άλλον. Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε ή εκ των ε, έξωθεν ε, προσπάθεια επιβολής διαπραγματεύσεων δεν οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, η οικονομία της χώρας είναι πολύ πιο ζωντανή από ό,τι οποτεδήποτε άλλοτε. Το Μογκαντήσου θα σας εκπλήξω με τις αναφορές που θα κάνω στο πόσο ζωντανή, ζωηρή είναι η οικονομία. Έχει επανέλθει το χρώμα, τα παιδιά τρέχουν στους δρόμους. Θαυμάσιο να βλέπει κανείς οικονομική δραστηριότητα. Πρόκειται για την επάνωδο της ομαλικής διασφορά, διασποράς, η οποία επενδύει. Αυτό λέει πολλά. Δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πραγματικό ζεστό χρήμα των Σομαλών. Και σε άλλες πόλεις διαπιστώνουμε το ίδιο φαινόμενο, αλλά κυρίως φαίνεται στο Μογκαντίσου. αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Μία από τις πραγματικές προκλήσεις για τη Σομαλία. Πρώτα απ' όλα, όπως ε, είμαι σίγουρος θα σας είπε και ο Πρόεδρος, η προτεραιότητά του είναι να υπάρξει περιβάλλον ασφάλειας. Αλλά ασφάλεια γι' αυτό δεν σημαίνει απλώς έλλειψη πολέμου σημαίνει να υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες. Δηλαδή χρειάζεται αστυνομία, δικαστικό σώμα. Οι πολίτες πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι το κράτος εγγυάται την ασφάλειά τους. Την καθημερινή ασφάλειά τους. Και βέβαια φυσικά τους προστατεύει και από απειλές τύπου Al-Shabaab. Αυτό παραμένει προτεραιότητα. Γι' αυτό οι διάφορες πολιτοφυλακές πρέπει να υπάρχουν σε ενιαία διοίκηση, πρέπει να εκπαιδευτούν από κοινού, να δημιουργηθεί πνεύμα σώματος σε οποιοδήποτε εθνικό σώμα ασφάλειας, όχι απλώς στον στρατό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει και μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Παίζει τον πρωτοπόρο ρόλο σε αυτό και θα συνεχίσει να έχει αυτόν τον ρόλο. Ε, δεν είναι μόνο η στήριξη που δίνουμε στην Αμισόμ, αλλά και το στρατιωτικό επιτελείο μας, με βάση και τις συνθήκες ασφαλείας, θα αναπτύξει μια επιχείρηση στη Σομαλία. Έχουμε το UCAP Nestor, που θα αναπτύξει την ασφάλεια στην ακτογραμμή. Θα βοηθήσει τη Σομαλία δηλαδή να δημιουργήσει ένα είδος ακτοφυλακής. Βασικό αυτό, η Αταλάντα συνεχίζει να λειτουργεί και έχει δραματικά μειωθεί η πειρατεία. Βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, πρέπει να είναι και κάτι ακόμη απόλυτα σαφές. Είναι πολύ εύθραυστη η κατάσταση. Όποιος ε, επαναπάβεται, κάνει σοβαρό λάθος και ο ίδιος ο λαός της Σομαλίας ε, σίγουρα το πιστεύει αυτό. Απλώς συγκρίνοντας με το παρελθόν πριν από ένα χρόνο έχουν υπάρξει ιδιαιτέρως ουσιώδης πρόοδοι. Δηλαδή ένα έθνος που έχει περάσει μέσα από αυτό το έρευος από το οποίο πέρασαν Σομαλοί κάποια στιγμή ένας τέτοιος λαός όπου υπόθη του λένε φτάνει, φτάνει αυτό το σκότος, θέλουμε να βγούμε στο φως, στον καθαρό αέρα, σε μια καλύτερη ζωή. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό, όλοι το καταλαβαίνετε, εφόσον ε, είστε πολιτικοί. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αριθμό. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε τη νέα πολιτική ηγεσία παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Αυτό θα επιτρέψει πρόσβαση για την ανθρωπιστική βοήθεια, ούτω ώστε όσοι είναι σε απελπιστική, απεγνωσμένη κατάσταση να λάβουν βοήθεια για να γίνουν και περαιτέρω επενδύσεις. Αν μπορούμε να αποκομίσουμε κάποια μαθήματα από τη Σομαλία για την υπόλοιπη περιφέρεια, θα μπορούσα να αφαιρθώ σε δύο-τρία πράγματα. Δεν λέω βέβαια ότι μπορούμε να κάνουμε άμεσε συγκρίσει. Πάντω μου κάνει εντύπωση το εξή. Η δέσμευση, προκειμένου να εγκατασταθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλεια, η δέσμευση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Και η δέσμευση τη Άμισομ έχει κλείσει πλέον τέσσερα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν δαπανηρή δεσμευσή αυτή, αλλά θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχή. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το ακόλουθο. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε πραγματικέ αφρικανικέ δυνάμει που έχουν καταφέρει να πετύχουν αυτό το τεράστιο επίτευγμα με σημαντικότατες θυσίε θυσίε αίματο, με φόρο αίματο, ουσιαστικά, από Αφρικανού προ του ομόεθνού του και προφανώς δεν πρόκειται για μια ανθρωπιστική ε, προσφορά. Θέλαν να αποφύγουν οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης, αλλά πραγματικά θα ήθελα να μιλήσω για τον επαγγελματισμό και την προσφορά τη σημαντικότητα της Άμισομ. Δεύτερον, Μπορεί να σταματήσουν οι διενέξεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα δύσκολο να καταφέρουμε να καθιδρύσουμε την ειρήνη. Και εδώ πέρα πάλι έχουμε μια σημαντική πρόκληση μπροστά μας όταν καταλαμβάνεται μία πόλη. Η δυνατότητα να έχουμε συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα τα οποία θα δώσουν συγκεκριμένε υποδομέ όπω κλινικέ, σχολεία, ένα σύστημα ίδρυυση. Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι θα πρέπει να κινούνται λίγο πιο γρήγορα. Και δεν αναφέρομαι απλώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρομαι στην γενικότερη διεθνή κοινότητα, στην ικανότητά τη να συντονίσει τι κινήσει τη και τι προμήθειε προκειμένου πραγματικά να ανταποκρίνονται στι πραγματικέ ανάγκε, είτε είναι πολιτικέ είτε είναι ανθρωπιστικέ. Νομίζω ότι ακόμα ψηλαφούμε, αν θέλετε, το πεδίο αυτό σε διάφορες χώρες που έχουν βρεθεί σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Ο τρίτο τομέα, στον οποίο θέλω να αναφερθώ να ακολουθώ, ουδέποτε θα επιληθούν τα προβλήματα μια χώρα, είτε πρόκειται για τη Σομαλία, είτε πρόκειται για κάποια άλλη, αν πραγματικά επικεντρωνόμαστε μόνο στη χώρα αυτή, απομονωμένα. Καταλαβαίνετε ότι όλε οι χώρε αυτέ έχουν και όμορε χώρε. Επομένω, το μελλοντική, η μελλοντική ασφάλεια της Σομαλίας εξαρτάται τελικά από το να αισθάνονται ασφαλείς και οι γείτονές της, από τη Σομαλία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ ε, ένα μεγάλο μέρος εργασίας μου έχει να κάνει με μια περιφερειακή παρουσία, δηλαδή να πηγαίνω από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα και να προσπαθώ ουσιαστικά να δημιουργήσω ένα δίκτυο εμπιστοσύνης ανάμεσα στις διαφορετικές πρωτεύουσε, στις διαφορετικές χώρες. Αυτό κάνω με την Αιθιοπία, με την Κένια, με το Τζιπουτί, που είναι όμορες χώρες και θα ήθελα να συνεργάζονται όλο και περισσότερο με το Μογκαντήσου. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Στο απότερο μέλλον επίσης η Σομαλία θα πρέπει να καταφέρει να μπει πάλι, να έχει μεγαλύτερη συνεργασία με τις εθνικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Σομαλία απλώς να δέχεται δάνεια. Θα πρέπει να καταφέρει να μπορεί να συμμετέχει επισήμως στην Παγκόσμια Τράπεζα, να μπορεί να δανείζεται από τους οργανισμούς αυτούς να μπορεί ουσιαστικά να λειτουργεί μακροοικονομικά. Προκειμένου όμω να γίνει κάτι τέτοιο, η Σομαλία θα πρέπει να έχει μια, ένα ανοιχτό σύστημα διαχείρισης, οικονομικής διαχείρισης, το οποίο να είναι επαγγελματικό, ανοιχτό, ευρύ. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο αυτό, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάποια σημαντικά γεγονότα στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώνει μία συνδιάσκεψη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ουσιαστικά θα κάνει πάρα πολλού ανθρώπου να αρχίσουν να στοχάζονται λίγο περισσότερο γύρω από το ζήτημα τη Ομαλία και τι πρέπει να γίνει. Το φθινόπωρο θα έχουμε και εμεί εδώ πέρα μία συνδιάσκεψη, η οποία θα καταλήξει ουσιαστικά σε μία συμφωνία ανάμεσα στη Σομαλία και τη διεθνή κοινότητα. Για να πω τα πράγματα με απλά λόγια αν η χώρα αυτή ουσιαστικά είναι κυρίαρχη τώρα και έχει κάποιες μελλοντικέ προοπτικές, αν πραγματικά θέλουμε να είναι ένας μελλοντικό μας εταίρος, ας πούμε ακριβώς πώς θα διαρθρωθεί αυτή η εταιρική σχέση. Ποιο θα είναι ο εταίρος μας, ποιο θα είναι το επιχειρηματικό μας πρόγραμμα, τι προπολογισμό θα έχουμε για αυτή την εταιρική σχέση, πώς θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τον προπολογισμό αυτό, όχι μόνο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα καταφέρει η ίδια η Σομαλία να δημιουργήσει ιδίους πόρους. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τη Σομαλία να σταθεί πραγματικά στα πόδια της. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, σε λιγότερα από τέσσερα χρόνια θα πρέπει να έχουν γενικές εκλογές σε όλη την επικράτεια της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, πολύ δύσκολος, αλλά προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Η χώρα αυτή πρέπει να σταθεί στα πόδια της και να καταφέρει να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο την πορεία της στο μέλλον. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτά όσον αφορά τη Σομαλία. Πολύ γρήγορα τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιους άλλους τόπους της περιοχής. Ερυθρέα. Είναι μια χώρα που πραγματικά έχει προσελκύσει την προσοχή σας, αλλά και τη δική μου την προσοχή. Έχω πάρει και τέσσερις φορές εκεί πέρα. Τον Ιανουάριο είχαμε κάποια επεισόδια στη χώρα, τα οποία παρουσιάστηκαν ως απομονωμένα επεισόδια και γεγονότα και φαίνεται τελικά ότι υπάρχουν όμως όλο και περισσότερα σωρευμένα, απομονωμένα γεγονότα και τέτοια επεισόδια στην Ερυθρέα. Και γύρονται κάποια ερωτήματα. Ουσιαστικά, μήπως ε, έχουν προκύψει κάποια ρήγματα, κάποιος κατακαιρματισμός ουσιαστικά στην εσωτερική οργάνωση της ιδιαίτερα απομονωμένης αυτής χώρας. Όπως ξέρετε, οι χώρες οι οποίες ε, καταλήγουν να είναι τόσο πονωμένε, έχουν και μια εσωτερική λογική για το πώ μπορούν να επιβιώσουν, πώ μπορούν να συνδιαλεγούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε μια φάση που είναι λογικό πλέον να ανησυχούμε για την Ερυθρέα. Όχι τόσο για το τι κάνει ή δεν κάνει η Ερυθρέα με τους γείτονές της. Η Ερυθρέα πραγματικά έχει λάβει πάρα πολλές κυρώσεις. Είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Το θέμα είναι τι κάνει η ίδια η χώρα στους πολίτες της και νομίζω ότι γύρονται κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Εγώ θα συνεχίσω να θέτω τα ερωτήματα αυτά κάθε φορά που πηγαίνω στη χώρα αυτή. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό εξετάζοντας την ευρύτερη περιοχή και όλους τους γείτονες να δούμε τελικά πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και βέβαια ξέρετε ότι η Αιθιοπία γνωρίζει τη χώρα αυτή καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα και οι Αιθίωπες είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως και οι υπόλοιποι γείτονες της ε, Ερυθρέας. Να σας πω το τελευταίο, το ακόλουθο για την Ερυθρέα. Πρόκειται για μια χώρα όπου ε, κάποιες περιοχές, οι οποίες ε, κατοικούνται κυρίως από μουσουλμάνους, σε σχέση με κάποια υψίπεδα τα οποία καλύπτονται από τους χριστιανούς βρίσκονται σε 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά στην Ερυθρά θάλασσα. Από την άλλη είναι η Εμένη. Καταλαβαίνετε ότι αν χάσει τον έλεγχο η χώρα αυτή αν γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση, τότε πραγματικά θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό επεισόδιο. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η εγκύτητα με την Ερυθρά θάλασσα. Θα ήθελα να το θέσω το ζήτημα αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τις ευθύνες μας, όχι μόνο η Ερυθρέα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Και ξέρετε ότι οι απειλές από την πειρατεία ουσιαστικά θα υπολείπονται, θα μοιάζουν ε, μηδαμινές μπροστά στον κίνδυνο τον οποίο μπορεί να δημιουργήσει στο μέλλον η Ερυθρέα. Σαφώς δεν έχω συγκεκριμένες απαντήσεις στο ζήτημα αυτό, πάντως θα ήθελα και τη δική σας συμβολή πώ μπορούμε να χειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια χώρα η οποία είναι τόσο απομονωμένη που έχει αρχίσει να παρουσιάζει τη δική τη ιδιαίτερη παθολογία, να το θέσω έτσι. Πώ μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. στι 21 Ιανουαρίου κάποιοι στρατιώτε πήγανε στην Ασμάρα και κατέλαβαν το Υπουργείο Πληροφοριών. Το γεγονό αυτό διήρκησε μία μέρα και όλο περιέργω δεν αντιλάγησαν πυροβολισμοί, δεν έγινε τίποτα. Στη συνέχεια υποχώρησαν, υπέβαλαν κάποια πολιτικά αιτήματα όσον ήταν κυρίω πολιτικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποχώρησαν στη συνέχεια. Μετά όμω από αυτό γίνανε πάρα πολλέ συλλήψει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στο επεισόδιο αυτό καθ' αυτό, αλλά και στα, στα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Ενδεχομένω να υπάρχει ένα άλλο υπόβαθρο δηλαδή πίσω από το μονομένο αυτό γεγονό. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι ο Νίλος. Εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Νείλος, να πω κάτι το οποίο προφανώς είναι σαφές σε όλους, αποτελεί την πηγή ζωής. Πηγή ζωής για πάρα πολλές χώρες. Για την Αίγυπτο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε 5.000 χρόνια ζωής και ταυτότητας, εθνικής ταυτότητας. Και όσο πιο νότια πηγαίνει κανείς στον Νείλο, τόσο συνειδητοποιεί ουσιαστικά τη συμβολή του ποταμού αυτού στην ζωή των γύρω περιοχών. Και ουσιαστικά έχουμε κάποια ζητήματα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Νείλου. Καταρχάς, τα τελευταία 30-40 χρόνια υπάρχουν όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής του Νείλου που φτάνει μέχρι τη λίμνη Βικτόρια, που ουσιαστικά έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον πληθυσμό τους. Ουσιαστικά θέλουν να καταφέρουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το νερό του Νείλου. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Η Αιθιοπία γνωρίζει ότι με την δημιουργία ενό φράγματο στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει υδροελεκτρική ενέργεια, πράγμα το οποίο θα καταστήσει τη χώρα αυτόνομη όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και θα τη επιτρέπει επίση να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στη γύρω περιοχή. Η Αίγυπτος ανησυχεί για όλε αυτέ τι νέε εξελίξει. Η ανησυχία την οποία θέλω τώρα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια περίπτωση η οποία μπορεί από τεχνικής φύσης, αν θέλετε, να επιληθεί. Υπάρχουν όλο και, περισσότεροι, όλο και περισσότερα πάθη τα οποία αναμοχλεύονται εξαιτία τη κατάσταση αυτή. Και αν τα πάθη αυτά ουσιαστικά πάρουν τον έλεγχο, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να δοθεί καμία απολύτω τεχνική λύση. Ουσιαστικά θα καταλήξουμε σε μια απόλυτη αναταραχή, σε ένα επικίνδυνο χάος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό σα λέω ότι θα πρέπει να δείξουμε απόλυτη ευθύνη, γιατί η Αιθιοπία και η Αίγυπτος είναι πολύ μεγάλε και σημαντικέ χώρε, οι οποίε συμβάλλουν ε, πάρα πολύ σημαντικά στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε δημιουργικού τρόπου για να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ και όλε τι υπόλοιπε ε, χώρε γύρω από τον Ήλο, προκειμένου να καταφέρουν να καταλήξουν σε μια κάποια λύση, σε μια βιώσιμη λύση για το πώς θα καταφέρουν να διαχειριστούν τα ύδατα του Νείλου. Πρόκειται λοιπόν για έναν τομέα τον οποίο όλο και περισσότερο εξετάζω. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω τώρα πολύ. Ας πάρουμε λίγο απόσταση από τα πράγματα. Άρχισα να μιλάω για την όλη αυτή περιφέρεια, για την όλη περιοχή. Αναφέρθηκα λίγο στην Κέννη, αλλά αν έχετε εσείς κάποιες ερωτήσεις ας μου τις υποβάλλετε βλέπουμε όλο και περισσότερο μια περιφέρεια η οποία περνάει από ένα μεταβατικό στάδιο. Μια περιφέρεια η οποία έχει τη δυνατότητα να αρχίσει ουσιαστικά να καταλαβαίνει πώ έχουν τα πράγματα. Βλέπουμε όλο και περισσότερου επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων που απευθύνονται σε μένα κάθε φορά που μιλάμε για ολοκλήρωση και μου έχουν πει ορισμένοι από αυτού, ωραία, σε καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε θεωρητικά τι θέλει να μα πει. Εσεί όμω έχετε την πραγματική έμπρακτη εμπειρία Βοήθησέ μας λοιπόν να καταλάβουμε πώς μπορούμε στην πράξη να πετύχουμε αυτή την ολοκλήρωση. Μη μας μιλάτε μόνο με θεωρητικά λόγια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι συναρπαστικό θα έλεγα, αλλά περιέχει και πάρα πολλές προκλήσεις. Για μένα αυτό είναι ο ουσιαστικός στόχος που έχουμε μπροστά μας. Βέβαια υπάρχουν ακόμα προκλήσει, ακόμα και κάποια εμπόδια, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να ξεπεράσουν τα εμπόδια του, να, καταφέρουν να ξεπεράσουν τι διμερεί διχόνοιε που υπάρχουν σε μια γεωγραφική περιφέρεια η οποία από ό,τι ε, φαίνεται έχει μια ιδιαίτερη παράδοση στον έρχεται σε διένεξη με τους γείτονές της παρά να συνεργάζεται με τους γείτονες. Και καταλαβαίνετε ότι το κόστος, το τίμημα είναι πάρα πολύ ψηλό. Πρέπει να ξεπεράσουμε πλέον την κατάσταση αυτή. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που μπορώ εγώ να δω είναι το ακόλουθο. Ότι ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα της ενέργειας στην περιοχή αυτή, με το πετρέλαιο και την υδροελεκτρική ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική και η οικονομική διάσταση της πολιτικής θα τροποποιηθεί πάρα πολύ. Θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να δούμε πώς μπορούμε από πολιτικής και οικονομικής πλευρά να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό. Πέρα από την ενέργεια έχουμε και το ζήτημα της θρησκείας καταλαβαίνετε ότι όλε αυτέ οι φυστάμενε διαφορέ τελικά περνάνε από τη θρησκεία. Είναι φιλετικέ, είναι θρησκευτικέ, είναι εθνοτικέ. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε όλε αυτέ τις διαφορές οι οποίε στην πράξη υφίστανται όμω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό ζήτημα, τι γίνεται στα πλαίσια του Ισλάμ στην Ανατολική Αφρική και γενικότερα στο κέρα τη Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι δεν αρκούν οι σύντομε επιφανειακέ περιγραφέ τη κατάσταση. Ξέρετε ότι ε, πολλές φορές ε, έχουμε κάποια φαινόμενα ριζοστικοποίησης του Ισλάμ σε κάποιες περιοχές, πέρα από το παραδοσιακό Ισλάμ που έχουμε στην Ανατολική Αφρική. Και βέβαια και η χριστιανική κοινότητα παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις και αντιδρά και αυτή με τη σειρά τη. Επομένω, δεν μιλάμε για μία μόνο θρησκεία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε πολλέ φορέ για την αντιπαράθεση και ουσιαστικά θα έχουμε όλο και περισσότερο μια κατάσταση στην οποία θα εμπλέκονται και πολιτικοί αλλά και θρησκευτικοί λόγοι. Θα πρέπει να αποφύγουμε όμως μια τέτοια διένεξη, μια τέτοια σύγκρουση. Θα πρέπει να έχουμε όμως τις παραμέτρους αυτές κατά νου. Ελπίζω πραγματικά να μην επαληθευτώ και ελπίζω ότι τελικά η ηρεμία και η ομαλότητα θα κυριαρχήσει στην περιοχή αυτή τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ολοκληρώσω στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι κάλυψα επαρκώς τα θέματα στα οποία πρέπει να αναφερθώ και ελπίζω ότι έχω προκαλέσει σε εσά παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ. Μας κάνατε μια παρουσίαση πολύ πλήρη από πλευράς γεωγραφικής. Από την πολιτική σκοπιά μας ε, δώσατε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις ε, στις οποίες εμβαθύνατε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι θέλουν το λόγο είτε για να αντιδράσουν είτε για να, είτε για να ζητήσουν περισσότερες διευκρινήσεις. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στο ρόλο της γειτονίας ως προς τη Σομαλία. Στο γεγονός ότι ο ρόλος των γειτονικών χωρών είναι καθοριστική σημασίας, ώστε να αντιλαμβανόμαστε αυτή τη χώρα όχι ως έναν εξαγωγέα αστάθειας να αλλάξει δηλαδή αυτή η νοοτροπία από πλευρά δική μα είναι πολύ σημαντικό για τη σταθεροποίηση αυτή, αυτή τη κατάσταση. Πέρα από την άμεση γειτονία όμω, ε, ενδεχομένως η Κένια και η Αιθιοπία πιο συχνά παρεμβαίνουν παρά σταθεροποιούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέραν από την άμεση γειτονία ε, επικρατεί η αίσθηση σύμφωνα με την οποία στη διεθνή κοινότητα όλοι οι μεγάλοι παράγοντες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση για τη σταθεροποίηση της χώρας αυτής ή μήπω ε, υπάρχουν υπόνοιες για κάποιες χώρες οι οποίες πέρα από την Ερυθρέα για την οποία γνωρίζουμε όλοι βεβαίως θα ήθελαν ή θα είχαν συμφέρον να διατηρηθεί ε, μια κάποιου είδους αστάθεια ή μπας περιπτώσει να μην ενθαρρύνουν τόσο σφόδρα την επιστροφή στην κανονικότητα και στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, ως προς τις ε, ευρωπαϊκές αποστολές οι οποίες αναπτύσσονται στο κέρας της Αφρικής. Η διάρθρωσή τους, η διασύνδεσή τους έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή, σας ικανοποιεί. Και αν όχι, ε, ποια σημεία επιδέχονται βελτιώσεων. Πιστεύετε και θεωρείτε ότι καλύπτουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της περιοχής, με την μέθοδο που ακολουθούμε ή λείπουν ε, και ε, θεμέλιες λύθη, αν θέλετε, από αυτό το οικοδόμημα που θέλουμε να χτίσουμε. Ο κύριος Γκάλερ και η κυρία Γκόμες στη συνέχεια. Κύριε Ρόντο, σας ευχαριστούμε θερμά για την ε, παρουσίασή σας, αλλά και για το γεγονός ότι έρχεστε στην υποεπιτροπή μας και μας ενημερώνετε τακτικά. Ως προς τη Σομαλία, ήθελα να θέσω διάφορα ερωτήματα. Καταρχάς, πώς ε, έχει διαμορφωθεί γενικότερα το κλίμα επιτόπου αποκομίζουμε την αίσθηση ότι σιγά αλλά σταθερά ο πληθυσμός αρχίζει και αποκτά εμπιστοσύνη στο νέο πρόσωπο της Σομαλίας, ότι είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα μείνει και θα παραμείνει και θα συνεχίζει να τη χάνει στήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Όταν προχωρούν τα στρατεύματα και καταλαμβάνουμε μία πόλη, ένα χωριό, διαδίδεται αυτή η φήμη ότι δηλαδή το κίνημα Al-Shabaab ε, έχει φύγει μια και καλή και θα προχωρήσουμε στην ανοικοδόμηση σχολείων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, ιατρικών υπηρεσιών. Το αξιολογεί ο κόσμος αυτό ως μια θετική έκβαση, ως μια πρόοδο. Ότι δηλαδή δεν εξυπηρετείται μια κάποια κρυφή ατζέντα. Δεν νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί κάποια στιγμή να επανέλθει ε, το κίνημα Al-Shabaab. Επομένως, ας μην προσυπογράψουμε με θέρμη αυτή τη νέα διοίκηση. Υπάρχει κάτι τέτοιο, αν όχι σε όλη τη χώρα, σε ορισμένα τμήματά της. Και από εκεί και πέρα. Βεβαίως και δεν μπορεί να εξαφανιστεί το Al-Shabaab κάπου θα βρίσκονται, παρόλο που οπισθοχωρούν. Ε, προς τα πού κατευθύνονται, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, έχουν πρόσβαση στη στήριξη που είχαν από τον οποιονδήποτε τους προσφέρει στήριξη. Και τέλος, η χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μέσου για την ειρήνη της Αμισόμ, της αποστολής της Ομαλία της Αφρικανικής Ένωσης. Πώς ε, διαγράφονται οι προοπτικές αυτές θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση στο ίδιο επίπεδο ή πρέπει να αναβαθμιστεί ή μπορεί ήδη να μειωθεί. Και τα ε, έθνη της Αφρικής που συνεισφέρουν έχουν ε, εκφράσει αυτό το πολιτικό μήνυμα ότι ναι θα συνεχίσουμε να στέλνουμε στρατεύματα για, την, ε, για το εγχείρημα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά κύριε Ρόντο που επισκέπτεστε την υποπιτροπή μας για άλλη μια φορά και για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και πληροφορίες που μας δώσατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Γκάλερ αναφέρθηκε στη Σομαλία και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω το εξής. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα πράγματα αναφέραμε στον πρόεδρο της Ομαλίας την εξής εξέλιξη. Ε, μια γυναίκα η οποία είχε βιαστεί βεβαίως απελευθερώθηκε στη συνέχεια, αλλά ο δημοσιογράφος που το δημοσίευσε συνεχίζει να είναι στη φυλακή. Οικοδομώντας τους θεσμούς ενός κράτους θα πρέπει να γίνεται σωστή δουλειά και θα πρέπει να υποβοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία για να υπάρξει σωστή ε, διακυβέρνηση, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι προφανές. Επομένως, σα ρωτώ, πώς, με ποιον τρόπο θα καταφέρετε να ε, διασυνδεθείτε όχι μόνο με την ΕΚΟ, ε, την υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και με το σκέλος το ανεπτεξιακό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε όποια βοήθεια δίδεται από πλευράς Ευρώπης να δίδεται για την υποστήριξη ε, και τη δημιουργία ε, σωστών ε, δομών και θεσμών διακυβέρνησης. Και ποιο ρόλο διαδραματίζει η Αφρικανική Ένωση εκτός από την Αμισόμ. Δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν, πιέζουν την κυβέρνηση της Ομαλίας να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα έθνη της Αφρικής Συν της άλλης, ένα ερώτημά μου έχει να κάνει με την Ερυθρέα. Ποιες είναι οι ιδέες σας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο απομονωμένο καθεστώς όσο αυτό που επικρατεί στην Ερυθρέα. Αυτό ρωτήσατε. Νομίζω εγώ προσωπικώς ότι έχουμε ένα εργαλείο το οποίο δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Σχεδόν. Και είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι δεν το χρησιμοποιούμε διότι πρόκειται για περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων. Ε, διαιτησία για την ε, σύγκρουση για τα σύνορα μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν παρέμενε ε, σιωπηρή. και η μόνη που δεν δέχτηκε τη διεθνή διαιτησία ήταν η Αιθιοπία για να μην ε, αποξενώσει και να δυσαρεστήσει τον Μάλες, ο οποίος όντως ήταν μια ε, κορυφαία προσωπικότητα στη χώρα. Ε, θα έλεγα ότι ήταν κορυφαίος και ως προς την ευφυΐα του, αλλά και ως προς το αδυσόπιτο του χαρακτήρα του. Κινούμενος πολύ κοντά στην απολυταρχική κυριαρχία. Ποτέ δεν ασκήσαμε πίεση ώστε να υπάρξει ε, συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βάσει της απόφασης που είχε ληφθεί. Και σε κάθε περίπτωση η Αιθιοπία ήταν αυτή η οποία δεν συμφώνησε. Νομίζω ότι έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει ένα εφαλτήριο για να ακουστεί ακόμα περισσότερο. Το λέω αυτό και γιατί θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον και της Αιθιοπίας, όχι μόνο της Ερυθρέας. Διότι έτσι θα εξασφαλίσει μία διόδο προς τη θάλασσα. Μέσω του ε, εντός εισαγωγικών τέκνου της που είναι η Ερυθρέα. Εγώ είμαι εξ αυτών που περιμένει τέτοιου είδου κινήματα όπως ε, τα κινήματα των στρατιωτών ε, να επιφέρουν την κατάρρευση του, της πολιτικής καθεστικής τάξης στην Ερυθρέα, η οποία είναι και μία από τις πιο δολοφονικές στην ευρύτερη ε, περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το θέμα έχει άμεση σχέση με την Αιθιοπία. Κάθε φορά που μιλάμε για την Ερυθρέα, έχει αυτό άμεση σχέση και με την Αιθιοπία οι μουσουλμάνοι όντως έχουν πολύ ε, στενούς δεσμούς με τους κατοίκους της Ιεμένης στην άλλη πλευρά της θάλασσας. Αυτό αφορά άμεσα ε, την Ερυθρέα προφανώς, αλλά αφορά και την Αιθιοπία. Γιατί το είδαμε και στη χώρα αυτή και τα τελευταία χρόνια ε, της θητείας του Μέλες, ο οποίος ουσιαστικά διατάραξε τις σχέσεις με την ε, μουσουλμανική κοινότητα και διατάραξε και τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, οι οποίες ήταν διατάρεκτες για αιώνες. Και εγώ όταν πήγα αυτό είδα, το 2008 αν δεν απατώ. Η κατάσταση των σχέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων επιδεινώθηκε ιδιαιτέρως έκτοτε και είχαμε και διαδηλώσεις της μουσουλμανικής κοινότητας διότι οι κρατικές αρχές παρενέβαιναν ε, στον ε, στη μουσουλμανική κοινότητα αυτή καθεαυτή. Και αυτό είναι αναπόφευκτο να έχει συνέπειες. Και μπορεί να έχει συνέπειες σαν και αυτές που αναφέρεται στην Ερυθρέα. Και θα ήθελα να πω ότι και εμείς κλείσαμε τα μάτια και κάναμε ότι δεν βλέπουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ως προς ε, την ε, ε, το καθεστώς στην Αιθιοπία και την αντιμετώπιση του κόσμου. Έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι είναι κρατούμενοι. Καταφέραμε να απελευθερωθούν δύο Σουηδοί δημοσιογράφοι, αλλά τι γίνεται με τους Αιθίωπες δημοσιογράφους. Ακόμα και ένας που έχει κερδίσει το βραβείο Πούλιτζερ συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή. Και τέλος, ως προς τον Νείλο, πράγματι οι επιπτώσεις και οι επιπλοκές με το Σουδάν είναι πολύ σημαντικές πώς αντιλαμβάνεστε την κατάσταση στο Βόρειο Σουδάν και με τον ε, ε ο Μαροσίν, τον πρόεδρο που έχει προσαχθεί στο Διεθνές ε, Δικαστήριο. Οι Κινέζοι υποτίθεται ότι θα, θα χτίσουν το φράγμα στην Αιθιοπία ή όχι. Και ποιο ρόλο διαδραματίζει η Κίνα, όχι μόνο σε, αυτές τις, σε αυτά τα σημεία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρουμε ποιο μονοπάτι κλασικό, ποια κλασική διαδρομή ακολουθεί η Κίνα αναζητώντας ε, ε, πόρους ε, πετρελαϊκούς, αλλά είναι ένα πρόβλημα ε, σοβαρό. Μπορείτε να τα αναπτύξετε όλα αυτά. Ο πρόεδρος διακόπτει. Αν θέλουμε ο Άλεξ να μας αναπτύξει τα θέματα αυτά, πρέπει να θέτουμε πιο σύντομες ερωτήσεις. Ο Ράινχαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ρόντο για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του. Μερικές, ε, μερικές ερωτήσεις μάλλον. Που σχετίζεται με την τελευταία παρουσίαση, ε, παρατήρηση της κυρίας Γκόμες. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Μέσω του Αταλάντα συνεργαζόμαστε με πολλούς άλλους ε, φορείς και, και διεθνείς και εθνικούς όπως η Κίνα. Τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι πέρα από την προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας. Δεύτερον, ορισμένοι και μεταξύ μας είναι μεγάλοι φίλοι της ανεξαρτησίας του Σομάλιλαντ. Όμως κατά πλειοψηφία συμφωνήσαμε ότι η επιδίωξη ενός τέτοιου στόχου θα είχε αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα για την περιοχή. Θα ήθελα να μας πείτε αν γίνονται τέτοιες αποσταθεροποιητικές προσπάθειες και μηχανογραφίες ή αν έχει κάπως ε, καλμάρει η κατάσταση. Τρίτον, οι Αμερικανοί έχουν χρησιμοποιήσει και ανεπάνδρωτα αεροσκάφη, drone στη Σομαλία. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε σε ποιο βαθμό και ε, τι άλλα μέσα χρησιμοποιούν. Υπάρχει συνεργασία στην αντιτρομοκρατική προσπάθεια μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Τέταρτον, στην εντολή της Αταλάντα συμπεριλαμβάνεται η προστασία των αλλιευμάτων της Σομαλίας και των περιοχών όπου γίνεται αλλία της Σομαλία έναντι τρίτων. Όμως, μέχρι στιγμής, η Σομαλία δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτό το καθήκον, να εκπληρώσει αυτό το καθήκον. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Τι δυνατότητες βλέπετε να υπάρχουν ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα απορρίπτονται και τοξικά απόβλητα στα ύδατα αυτά. Αναφερθήκατε στην έκκληση που απευθύνθηκε σε εσά, μιλήστε μας. Έχετε επαρκές προσωπικό επαρκείς πόρους, επαρκή στήριξη μέσω των ευρωπαϊκών δομών για να το κάνετε αυτό. Μήπως χρειάζεστε περισσότερο προσωπικό, περισσότερη βοήθεια για να επιτύχετε στην εργασία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Αλέξανδρε, ίσως να χρειαστεί να υπερβείς λίγο το χρόνο. Σας ευχαριστώ όλους. Για να τα δούμε με τη σειρά. Η αρχική ερώτησή σου, Αρνό, ήταν ε, ποιες είναι οι απόψεις μου στην ουσία για την περιοχή του κόλπου. Θα δούμε και τα άλλα. Κοίταξε, ο κόλπος της Αφρικής, γύρω από τη Σομαλία και στο Τζιμπουτί, θεωρεί ότι είναι επέκταση του κόλπου όπως είναι όλη η Ποσαχάρη Αφρική. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορική πραγματικότητα. Εκεί αναπτύχθηκε η διάδοση των ε, θρησκειών. Λογική αυτή η σχέση. Γιατί και ατύπως ε, έτσι γίνεται το εμπόριο. Είναι βεβαίως και νόμιμο και παράνομο. Είναι και εμπορία ανθρώπων, όπλα, ναρκωτικά, τα πάντα. Είναι προς το συμφέρον λοιπόν όλων να διασφαλίσουμε ότι όλη αυτή η περιοχή λαμβάνεται υπόψη μαζί με τον κόλπο. Έτσι τα σκέφτομαι εγώ. Δεν θα ήταν σωστό στρατιωτικά, διπλωματικά να επιχειρήσεις να κάνεις κάτι για την περιοχή χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ευρύτερη περιοχή. Βεβαίω τώρα Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά με τις χώρες αυτές. Πολύ σοβαρά. Γιατί μπορούν να συμβάλλουν και πραγματικά είναι προς το συμφέρον τους. Να σταθεροποιηθεί η περιοχή σίγουρα εμπορικά, αλλά και για λόγους ασφάλειας. Αλλά εκτός από αυτό και παράλληλα, αν πρόκειται να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές, δεν θέλουμε να είναι σαν και εμάς. Αλλά εάν έχουν ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως ε, επενδυτικές τράπεζες που λειτουργούν διεθνώς, τότε και οι επενδύσεις του στη Σομαλία, η βοήθεια στη Σομαλία πρέπει να γίνονται με το βαθμό διαφάνειας που ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη εντός της Ένωσης. Εδώ υπάρχει ακόμη μια διαφορά φάσης μεταξύ ημών και κάποιων από τις χώρες αυτές. Και αυτό θέτει την Ένωση ενώπιον μια σημαντικής πρόκλησης. Η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από άλλες χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι θέμα που πάντα μας απασχολεί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θέτουμε κάποια πρότυπα που άλλοι υπονομεύουν. Αλλά Υπάρχει και ένα στρατηγικό θέμα, σημαντικό. Θα ήταν όχι μόνο για μας, αλλά και για τους πολίτες της περιοχής, πολύ επικίνδυνο, η περιοχή να γίνει χώρος ανταγωνισμού επιρροών θρησκευτικών. Έχει υπάρξει ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίω ω ένα βαθμό συμμερίζομαι Άννα την άποψή σου για την Αιθιοπία, αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα. Η ακτή Σουαχίλη της Ανατολικής Αφρικής που υπήρχε όταν μεγάλωνα είναι πολύ διαφορετική. Τα τζαμιά δίπλα στα οποία μεγάλωσα τώρα λένε άλλα τροπάρια. Θα πρέπει να δούμε τι έγινε, γιατί και πού το πάει η κατάσταση. Οπότε περνάμε, αυτό μας φέρνει φυσιολογικά στην ερώτηση του Σουδάν. Στο θέμα του Σουδάν. Εκεί οι μουσουλμανικές ελίτ της περιοχής και ακόμη και στην Δυτική Αφρική εκεί εκπαιδεύονται. Δεκαετίες τώρα στο Σουδάν. Κάτι γίνεται. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε πολύ καλύτερα. Αν θέλουμε να εξαγάγουμε βάσιμα συμπεράσματα. Για τον κόλπο λοιπόν, Για τον κόλπο έλεγα δεν είναι θέμα γένειας. Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς για το ποια είναι τα συμφέροντά μας όταν συζητάμε με άλλους. Και όταν συζητάμε με χώρες του κόλπου, είναι καλό να πάμε και να μιλήσουμε ανοιχτά. Γιατί στην τελευταία ανάλυση, αν ο κόλπος θέλει να επηρεάσει, ας πούμε, τη Σομαλία, σας διαβεβαιώ ότι και οι γείτονε, οι διπλανοί θα αντιδράσουν. Και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανένας. Η άλλη χώρα που έχει παίξει ένα πολύ προβεβλημένο ρόλο είναι η Τουρκία που τα τελευταία ένα-δύο χρόνια έχει μπει στην περιοχή, έχει κάνει πολύ θεαματικές ενέργειες με υψηλή ορατότητα. Συμβάλλει βέβαια, αλλά είναι ασήμαντα τα ποσά με τα οποία συμβάλλει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι των ποσών Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τους πούμε να συμπεριφερθούν όπως όλοι οι εταίροι. Να καθίσουμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε τις ιδέες μας και να δούμε τι πρέπει να εφαρμόσουμε, τι είναι εφικτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώ τώρα το να επιχειρεί ο καθένα να κάνει μόνο του κάτι, τελικά ε, καθίσταται τμήμα του προβλήματο και όχι τη λύση. Οι αποστολέ τη Ένωση. Αν το δούμε με ιστορική προοπτική και ξέρετε εγώ μόνο 15 μήνες ασχολούμαι με αυτή την περιοχή πολλές έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα Τι διαπιστώνω Κάθε αποστολή προσπαθούσε να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη Άμισομ, Αταλάντα μετά το EUTM μετά τον Έστορ Έτσι γίνεται παντού. Σύνηθε φαινόμενο. ιδίω ε, για θέματα ασφάλεια. Το έχουμε δει και σε πολλέ άλλε περιοχέ. Αλλά σε κάποια φάση πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Πώς το κάθε μέσο ενεργεί επί του εδάφους. Επί τόπου δηλαδή. Και επίσης ε, να τα κατανείμουμε και γεωγραφικά. Κατά το τελευταίο δεκάμινο η Σομαλία έχει γίνει πολύ πιο προσβάσιμη. Άρα λογικό είναι η καταπολέμηση της πειρατείας ας πούμε να γίνεται στο μέτρο του δυνατού από τη Σομαλία, να βασίζεται στη Σομαλία. Αυτή είναι μια μόνιμη συζήτηση μεταξύ υπηρεσιών. Πώς να δημιουργήσουμε συντονισμό των δράσεών μας. πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρές αποτιμήσεις της κατάστασης ασφαλείας του προσωπικού. Να προστατεύουμε το προσωπικό μας επιτόπου. Και εδώ λογικό είναι να λένε πολλοί δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο το προσωπικό μας. Αλλά αν δεν το κάνουμε, κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι επιτακτικοί οι λόγοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή χρειάζεται θάρρος. Γιατί το θάρρος έχει πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά αποτελέσματα. Ξέρετε, είναι σαν να κάνει υπασία. Το άλογο ξέρει αν φοβάται ο αναβάτης και τον πετάει. Αλλά από τη στιγμή που θα τους δείξουμε, που θα δείξουμε ας πούμε στον ύπο ότι είμαστε κύριοι του, τότε θα καλπάσουμε. Είναι λοιπόν ε, πολύ ευαίσθητη περιοχή αλλά και ευαίσθητα αυτά που προτείνω. Γιατί προτείνω λοιπόν να διατρέξουμε κινδύνους. Και δεν είμαι στρατιωτικός, να είναι σαφές. Αλλά υπάρχει μια πολιτική κινητικότητα που το θάρρος θα μπορούσε να επιτύχει πολλά σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη συγκυρία. Οι Σομαλοί περιμένουν πολλά από εμά. Να αναρωτηθούμε λοιπόν όσο λιγότερα κάνουμε τόσο μεγαλύτερο κενό θα υπάρξει και το κενό αυτό κάποιος άλλος θα το καλύψει. Άρα ερχόμαστε στην ερώτηση, Μάικλ, που έθεσες. Ε, εμπιστοσύνη, ανοικοδόμηση, σταθεροποίηση. Μην ανησυχείτε για διάφορες φήμες. Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Καταλαβαίνω. Αλλά τι εννοώ. Καλές είναι οι φήμες. Αλλά πρέπει οι φήμες να ακολουθούνται από συγκεκριμένη δράση και παροχή υπηρεσιών. Σε αυτή τη φάση λέμε πολλά για την σταθεροποίηση. Ενδιαφέρουσα λέξη. Σταθεροποίηση, σταματάνε οι συγκρούσεις, ε, ε, απελευθερώνεται μια πόλη και πάμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σταθερή κατάσταση. Αλλά για πολλούς η σταθεροποίηση είναι κακή έννοια. Γιατί αυτό σημαίνει συνεργασία με κάποιες πολιτοφυλακές και άρα υπάρχουν προβλήματα για τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των διοικήσεων που δημιουργούνται κτλ. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ πρακτικό θέμα. Αφαιρούμε μια πόλη από τον έλεγχο του Σαμπάμπ. Χρειάζεται σχολείο, χρειάζεται δικαστήριο, κλινική, πόσιμο νερό κτλ. 100.000, 200.000 ευρώ. Αρκούν για να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Ωραία. Αλλά δεν υπάρχουν οι φορείς για να προχωρήσουν στην οικοδόμηση αυτών των εγκαταστάσεων. Αυτό πρέπει να γίνει και πολύ γρήγορα. Και γίνονται προσπάθειες. Έχουμε τώρα αυτό το περιθώριο, αν μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε για να σημειωθεί πρόοδος, τόσο το καλύτερο. Και ένα πράγμα έχω στο μυαλό μου. Σέβομαι πλήρως ε, τις ανησυχίες ε, των αρμοδίων για ανθρωπιστικά θέματα, για κάποιες τέτοιου τύπου εργασίες, αλλά πρέπει να την κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά και ούτω ή άλλω ε, τι πρώτε εβδομάδε, πρώτου μήνε, ο στρατό που έχει απελευθερώσει και που κατέχει την περιοχή κάνει αυτέ τι δουλειέ. Όσο περισσότερο προχωράνε αυτέ τι δουλειέ, αυξάνεται η ασφάλεια, δημιουργείται θετικό κλίμα και άλλοι λοιπόν φορεί μπορούν και αυτοί να μπουν και να αρχίσουν να εργάζονται. Πάντα βέβαια προσπαθούμε να ανακτήσουμε τις καθυστερήσεις σε αυτό το τομέα όσον αφορά την Al-Shabaab, πώς έχει κατάσταση, πού βρίσκονται. Ίσως πουθενά αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει την τακτική τους. Κάθε φορά υποχωρούν συστηματικά, καθώς βλέπουν ε, τις δυνάμεις της Άμισομ να φτάνουν ή ε, άλλες ε, στρατιωτικές οργανώσεις από τη Σομαλία. Έχουν πάει κάπως προς την επαρχία, προς την Ήπεθρο από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί Σαμπάμπ οι οποίοι καταλείπουν πλέον την οργάνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά πηγαίνουν στην Άμισομ και υπάρχουν μάλιστα και κάποια ειδικά προγράμματα ενσωμάτωσή του, τα οποία δημιουργούνται και πρέπει να δημιουργούνται. Ο σκληρό πυρήνα όμω παραμένει. Παραμένει σκληρό πυρήνα τη οργάνωση. Ξέρω ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη τη Al Shabaab, μέλη που ας το πούμε ότι ε, συνάδουν ουσιαστικά η νοτροπία του συνάδει με την νοτροπία της βασικής κυβέρνησης. Σιγά σιγά αυτοί, όντας συνοδοιπόροι, μπορούν να έρθουν με το μέρος της κυβέρνησης. Και αργά ή γρήγορα πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Ουσιαστικά έχουμε κάποιες εκατοντάδες οι οποίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα. Και δεν αναφέρομαι καν σε εκπροσώπου τη Τζιχάντα αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν φύγει πλέον γιατί συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα πλέον στην ε, Σομαλία. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι κάνει ο σκληρό πυρήνα, ποιοι είναι οι στόχοι του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εμποδίσουμε οποιαδήποτε επέκτασή του προ άλλε περιοχέ πέρα από τη Σομαλία. Και στη συνέχεια θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε μετακίνησή τους προς την Πούντλαντ ή τη Σομάλιλαντ. Ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές έχουν εκεί πέρα βασικά εισοδήματα. Τώρα, όσον αφορά την ε, διευκόλυνση το μέσο για την ειρήνευση. Ναι, σημαντικό αυτό αρκεί να μπορούμε να το χρηματοδοτούμε. Και ξέρω ότι η απόφαση αυτή είναι πολύ δύσκολη, αλλά πρέπει να ληφθεί γιατί είναι σημαντικό το μέσο αυτό. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τώρα αυτόν τον αγώνα, ενώ σιγά σιγά τον κερδίζουμε τελικά. Αυτό θα είναι μια απόλυτη τραγωδία και θα στείλει το χειρότερο δυνατό μήνυμα προς τα έξω σε μια περιφέρεια που ουσιαστικά έχει να κερδίσει πάρα πολύ από το μέσο αυτό και που ουσιαστικά εμείς την χρειαζόμαστε. Την χρειαζόμαστε σταθερή. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε με το μέσο αυτό, αρκεί βέβαια και άμυσο να μπορεί να συνεχίσει τη δράση της, αλλά θα πρέπει να έχει βαθμιαία ένα μικρότερο ρόλο, όσο σιγά σιγά θα αυξάνονται οι στρατιωτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας. Στα πλαίσια όλου του έργου που λαμβάνει η χώρα στη Σομαλία έχουμε και προγράμματα επιβολής του κράτους δικαίου. Πολύ σημαντικά προγράμματα για τα οποία εμείς είμαστε οι πιο σημαντικοί χρηματοδότες μαζί με τα Ενωμένα Έθνη και νομίζω πλέον ότι αρχίζουμε να φεύγουμε και από τη Μογκαντήσου, δεν επικεντρώνονται μόνο και πέρα τα προγράμματα, αλλά πηγαίνουν και προς την Ήπεθρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά για το κράτος δικαίου, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε και ένα δικαστικό σύστημα, να έχουμε μία εκπαίδευση, αν θέλετε, δικαστών σε μία χώρα από την οποία οι δικαστές απουσίαζαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η Αφρικανική Ένωση έχει και αυτή ένα ρόλο, αλλά είναι πιο πολιτικός ο ρόλος αυτός αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα την Ερυθρέα. Μάλλον, ας παραμείνω μια στιγμή στην Σομαλία, πρωτού προχωρήσω σε άλλες περιοχές. Σομάλιλαντ. Ξέρετε τώρα ότι μετά από 20 χρόνια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που προσπαθούμε να ενώσουμε πάλι μια χώρα η οποία είχε κατακαιρματιστεί. Η απόπειρα αυτή τη στιγμή να νομιμοποιήσουμε την αυτονομία ενός τμήματος της χώρας αυτής ουσιαστικά θα στείλει ένα εντελώς λαθασμένο μήνυμα και βλέπω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής αυτής του Σομάλι Λάντ δεν ζητούν αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Δεν πηγαίνουν από εδώ και από εκεί ζητώντα αυτονομία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται κάποιε πολύ σοβαρέ όριμες συζητήσει, ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Σομαλία. Το θέμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά κατά την άποψή μου, η δική μου αν θέλετε προσωπική άποψη, είναι η ακόλουθη. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε τώρα με το ζήτημα αυτό. Α αφήσουμε καταρχά του ίδιους του ομαλού να επιλύσουν το ζήτημα αυτό. Να δούνε ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Διεξάγονται πάρα πολλέ συζητήσει αυτή τη στιγμή. Και του εύχομαι, εύχομαι καλή επιτυχία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που ήδη εμπλέκονται στι εσωτερικέ αυτέ συζητήσει Και δεν αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στο καθεστώ. Δεν εύχομαι μία έκβαση, τη μία την άλλη έκβαση για το καθεστώ. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η μεταξύ του συνεργασία. Για την Αταλάντα τώρα. Αν κατάλαβα την ερώτησή σας για τα ζητήματα κατά της πειρατείας. Προφανώς οι περισσότεροι συμφωνούμε με όλες αυτές τις δράσεις κατά της πειρατείας. Όλοι εμπλέκονται με τον ένα τον άλλο τρόπο, οι χώρες του κόλπου αλλά και πιο πέρα από τον κόλπο και βλέπω ότι θα συνεχιστεί αυτό στο μέλλον. Φτάνουμε όμως σε ένα πολύ ενδιαφέρον στάδιο πλέον. Στάδιο στο οποίο δεν θα πρέπει απλώς να μας απασχολεί μόνο η υπάταξη της πειρατεία, που νομίζω ότι σε αυτό ουσιαστικά αναφερθήκατε και στο, στο ερώτημά σας, θα πρέπει ουσιαστικά να δούμε ότι ο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό, ο οποίο πηγαίνει από την Ινδία και το Πακιστάν, από το κόλπο του Άντεν μέχρι τη Μαδαγασκάρη, φανταστείτε όλη αυτή τη γεωγραφική ζώνη, είναι μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει ουσιαστικά αστυνόμευση όσον αφορά τα ανοιχτά, την ανοιχτή θάλασσα και ουσιαστικά συμβαίνουν πολλά και επικίνδυνα πράγματα. Μα ανησυχεί σαφώ η πειρατεία, αλλά έχετε ασχοληθεί καθόλου με τη διακίνηση των ναρκωτικών που έρχονται από το Πακιστάν προς την Ανατολική Αφρική. Ελάχιστοι αναφέρονται στο ζήτημα αυτό. Αλλά ουσιαστικά αυτό παρεμποδίζει την ίδια την αφρικανική ζωή και πολιτική ενδεχομένω να μην βλέπουμε τα αποτελέσματα όσο άμεσα τα βλέπουμε με την πειρατεία, αλλά υπάρχουν επιπτώσει και από τη διακίνηση ναρκωτικών. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα τα οποία σφαιρικά θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Θα πρέπει σαφώ να δούμε τι έχει κάνει η Αταλάντα, τι συνεχίζει και κάνει η Αταλάντα και την αλληλεία πρέπει να προστατεύσουμε. Ξέρετε όμω ότι ε, υπάρχει μια αποκλειστική ε, ζώνη για την ε, Σομαλία και θα πρέπει να αναπτυχθεί. Α, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μα απασχολήσουν μόνο κάποια εκατοντάδε μίλια πέρα από την ακτή τη Σομαλία, θα πρέπει να δούμε ακόμα και πιο πέρα, ακόμα πιο ανοιχτά, τι ακριβώ γίνεται. Ποια ζητήματα υφίστανται. 50 κιλά ηρωίνη ξέρετε ότι μπορούν να έχουν πολύ οδυνηρέ επιπτώσει, όχι μόνο στην ανθρώπινη υγεία, αλλά σε ολόκληρε χώρε και περιοχέ. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ευρύτερο ερώτημα το οποίο ε, ουσιαστικά θα πρέπει να απαντηθεί. Όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Ξέρετε, πολλές φορές ότι μέσα στο Μογκαντήσου τα οι παδρομένα αεροσκάφη τα οποία πετάνε. Δεν υπάρχει μια επίσημη συνεργασία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια προγράμματα κατά τη θερμοκρατίας τα οποία εφίστανται. Παράλληλα όμω, εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούμε περισσότερο μια ευρύτερη στρατηγική για να δημιουργηθεί ένα τομέα ασφαλείας για την ίδια τη Σομαλία και επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην πολιτική αναπτυξιακή πτυχή πολύ γρήγορα να απαντήσω και στα ζητήματα τα οποία ακούστηκαν για την Ερυτρέα. Έχετε δίκιο. Μπατ μεν υφίσταται, αλλά δεν είναι μόνο Δεν νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει μόνο το ζήτημα αυτό στο οποίο επικεντρωθήκατε, αλλά θα πρέπει περισσότερο να δούμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην Ερυτρέα και την Αιθιοπία. Είναι δύσκολο να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σαφώς θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για το σνοριακό ζήτημα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω κάτι για την Ερυθρέα. Πάντως, τουλάχιστον για την Αιθιοπία, νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια βούληση προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Και είναι προφανώς προς το συμφέρον τους, όπως το είπατε κι εσείς. Και είναι οι πρώτοι άλλωστε που τον αναγνωρίζουν αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει πίεση μέχρι ενός σημείου. Αλλά η μόχλευση αυτή είναι δύσκολο πολλές φορές να αξιολογηθεί. Όσο περισσότερο μιλάμε πάντως με τα εμπλεκόμενα μέρη, τόσο περισσότεροι τρόποι συνεργασίας τελικά βρίσκονται στο τέλος. Αναφερθήκαμε στο ζήτημα της Αιθιοπίας και του μουσουλμανικού πληθυσμού και πραγματικά μην επικεντρώνεστε μόνο σε αυτό. Υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα στην περιοχή το οποίο πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλύτερα και ενδεχομένω ε, να επηρεάζει όλη την περιοχή από το Σαχέλ πηγαίνοντα προ τα Ανατολικά. Σε όλο αυτό το τόξο, όλο αυτό το τόξο πρέπει να μα απασχολήσει. Για το Σουδάν τώρα. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Να σας διορθώσω σε κάτι. Το φράγμα στην Αιθιοπία δεν το χτίζουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι δεν εμπλέκονται καθόλου σε αυτό. Χτίζεται με χρήματα, μάλλον η χρηματοδότηση είναι καθαρά αιθιοπική χτίζεται πραγματικά από χρήματα που προέρχονται από τους Αιθίωπες. Δεν εμπλέκονται οι Κινέζοι. Καθόλου. Όσον αφορά τώρα το Σουδάν. Δεν έχω πάει Έχουμε έναν ειδικό εντεταλμένο, ο οποίος είναι αρμόδιος για ζητήματα του Σουδάν. Με την συνάδελφο αυτή θα πρέπει να συνομιλήσετε περισσότερο. Προφανώς συνεργαζόμαστε, αλλά αυτή είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από μένα να σας μιλήσει για το Σουδάν. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω με ακρίβεια για το Σουδάν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι καλύψαμε ε, όλα τα ερωτήματα τα οποία ακούστηκαν. Πολλά πράγματα ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε τακτική πάντως ανταλλαγή απόψεων και θα έχουμε και στο μέλλον και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα για μερικά λεπτά. Την Προεδρία θα την αλάβει ο Κριστόφ για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ.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 Ladies and gentlemen, we will start in... Θα ξεκινήσουμε σε δύο λεπτά. Περιμένουμε την κυρία Λόιζιν. Ladies and Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε. Πολλά μέλη της Επιτροπής μου είπαν ότι βιάζονται. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να επιταχύνουμε το ρυθμό μας. Θα ασχοληθούμε με το σχέδιο έκθεσης για τις εξαγωγές όπλων στο πλαίσιο της κοινή θέσης. Η κυρία Λόεζιν είναι η συγγήτρια μας παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης το Φεβρουάριο και σήμερα το εξετάζουμε αυτό για δεύτερη φορά. Υπάρχουν ήδη τροπολογίες. 175 αν δεν απατώμε, για τη και σκιώδη Έχετε το λόγο, κυρία Λέζιν, για πέντε λεπτά. <coughs> Ίσως θα χρειαστώ λίγο περισσότερο γιατί βήχω και θα κάνω πολλές διακοπές. Ε, με συγχωρείτε, αλλά θα χρειαστεί να βήξω ορισμένες φορές. Ευχαριστώ λοιπόν. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις πολλές και σχεδόν αποκλειστικά συμπληρωματικές και ε, επικοδομητικές τροπολογίες. Να συνοψίσω την έκθεση λοιπόν. Επιδιώκουμε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ενημέρωση και ε, πιο εναρμονισμένη και ε, ρωμαλαία εφαρμογή. Θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε, όπως κάνουν ορισμένοι συνάδελφοι, να ε, μειώσουμε την ε, ένταση της έκθεσης αυτής. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξη γιατί μπορώ να κάνω κάποια σχόλια και κάποιες συμβαστικές προτάσεις για τις τροπολογίες. Για την αιτιολογική σκέψη F και την τροπολογία 25 και 26 δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα για να ε, πάρουμε την ακριβή διατύπωση του άρθρου 10 της κοινής θέσης για την ε, έλλειψη ενός καταλόγου ε, για την αιτιολογική έσκεψη F. Συμφωνώ με την πρόταση ΜΕΚη και ΤΕΡΟ γιατί γράφουν ότι αυτό είναι μια διαπίστωση και δεν αποτελεί απέτηση. Ίσως θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια διατύπωση όπως την τροπολογία 32. Οι τροπολογίες 31 και 39 τροπολο, ε, μετατρέπουν, μεταβάλλουν την έννοια των αιτιολογικών σκέψεων και τροπολογία 40 νομίζω ότι προτείνει μία απάλληψη που δεν είναι τελογημένη γιατί ναι μεν δεν είναι ικανοποιητική η κοινή θέση αλλά περισσότερη πληροφόρηση υπάρχει χωρίς αυτή. Οι επόμενες μέχρι την τροπολογία 250 είναι όλες πολύ επικοδομητικές, οπότε για μένα είναι απόλυτα αποδεκτές. Η τροπολογία 57, κατά τη γνώμη μου, ε, περικόπτει κατά πολύ την ε, ε, περιγραφή των εξαγωγών όπλων προς την Λιβύη, ούτως ώστε να μην έχει έννοια. Κανένας δεν έχει αναφέρει κάτι που να τροποποιεί αυτή την πολύ καλή ε, περιγραφή παραδείγματος. Συμφωνώ με την κυρία Νικολά και την κυρία Κρόνμπεργκ, εάν η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο, στην περιοχη ΜΕΝΑ M1 λαμβάνεται υπόψη και γι' αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να γίνουν καθόλου ε, εξαγωγές όπλων. Η τροπολογία για την κοινωνία των πολιτών ε, με βρίσκει σύμφωνη για την τροπολογία 65 συμφωνώ προς το παρόν, αλλά θα ήθελα να τη συμπληρώσω προφορικά, ούτως ώστε να αναφέρουμε τα νέα στοιχεία από το Ινστιτούτο για την Ειρήνη Σύπρη, όπου λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο δεύτερος εξαγωγέας όπλων. Παράγραφος 2 τώρα και οι τροπολογίες που την αφορούν θα μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβασμό που να ανταποκρίνεται στο, στο πνεύμα των τροπολογιών 66-72 για την παράγραφο 3 και ιδιαίτερα την τροπολογία 79 της κυρίας Κοπά. Την υποστηρίζω. Όπως και η κυρία Κοπά, συμφωνώ με την περιγραφή της κατάστασης. και επεξηγεί και τη δική μου τροπολογία για το ίδιο σημείο, την ίδια παράγραφο. Πιστεύω ότι και εδώ θα βρούμε μια συμβαστική λύση για τις τροπολογίες της παραγράφου 4. Θεωρώ ότι με βάση τροπολογίες 81 και 82 μπορούμε να βρούμε συμβασμό. Για τις τροπολογίες 84 και 85 Από τότε που εκπονήθηκε η έκθεση έχω συζητήσει με διάφορες ε, ε οργανώσεις και έχω μάθει ότι ε, οι εξαγωγές όπλων και η έλλειψη πληροφόρηση για το πώς γίνονται, πού πάνε και σε ποιον και λόγω της ε, μη επαρκούς εφαρμογής των κανόνων. Υπάρχουν πολλές μελέτες γι' αυτό και μια εναρμονισμένη εφαρμογή της κοινή θέση θα ήταν αναγκαία. Λυπάμαι που οι τροπολογίες δεν προτείνουν ε, κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της κοινή θέσης. Αλλά πιστεύω ότι με βάση αυτές τις τροπολογίες θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Για την παράγραφο 10 θα επιδιώξω συμβιβασμό με βάση τις τροπολογίες 114-116 και ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία γι' αυτό. Για την παράγραφο 14 και το αίτημα για περισσότερη πληροφόρηση. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες 124-127 είναι δυνατόν να αποτελέσουν βάση ικανοποιητικού συμβασμού. Για το ΑΤΤ δεν βλέπω να υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις και χαίρομαι γι' αυτό. Και χαιρετίζω αυτή την συμπλήρωση. Μπορώ να την ε, συμπεριλάβω. Παρατηρώ ότι διαφορετικές περιγραφές καθώς και κάποια γλωσσικά θέματα ε, έχουν να κάνουν ακριβώς με τη μετάφραση. Όλοι για το θέμα της μετατροπής φαίνεται να συμφωνούν, αλλά αυτό το ανέμενα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να υπάρξουν ε, επικοδομητικοί συμβιβασμοί. Κατόπιν, τις επόμενες μέρες, θα υποβάλουμε ε, μέσω email συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα με χαρά να δώσω το λόγο στον εαυτό μου, γιατί είμαι σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚΑ. Dziękuję bardzo pani, pani poseł Luizing za gotowość do kompromisu. My dzisiaj omawialiśmy na... E, Και θα ήθελα να πω ότι σήμερα στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση της ομάδας μας συζητήσαμε την έκθεση αυτή. Δεν πρόκειται λοιπόν να εμβαθύνουμε τόσο στις τροπολογίες. Δεν πρόκειται να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, διότι σήμερα στις 9.30 το πρωί λάβαμε το μεταφρασμένο κείμενο και άρα δεν είχαμε χρόνο να διαβάσουμε όλες τις τροπολογίες. από τη στιγμή που είχαμε και συνεδρίαση στην Επιτροπή αργότερα. Σε γενικές γραμμές όμως θέλω να σας πω το εξής. Η συζήτηση που κάναμε έδειξε ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης και ελπίζω σε ανταλλαγή μηνυμάτων με την κυρία Βουλευτή και αν θέλετε να συναντηθούμε συναντιόμαστε επίσης. Δύο μερικά σχόλια θα ήθελα να κάνω. Ως ομάδα νομίζουμε ότι δεν θα ήταν δίκαια ε, τόσο η ρύθμιση αυτή, η νομοθετική. Γιατί? Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος να πλήξει αυτό τον ε, ε, ευρωπαϊκό κλάδο άμυνας. Και γι' αυτό υποβάλαμε αυτές τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις στον τομέα της ασφάλειας και με τις θέσεις εργασίας. Άλλωστε, χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται σε αυτό το κλάδο στην Ευρώπη. Επομένως, αυτό είναι και το πνεύμα των τροπολογιών μας, ε, τις οποίες σας έχουμε υποβάλει και φαντάζομαι ότι τις ε, γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα, ήθελα να πω και το εξής. Πολλές τροπολογίες και δικές μας, αλλά και από άλλες πολιτικές ομάδες υπάρχουν και αναφέρονται στο εδάφιο 27. Θα έλεγα και για πολύ σοβαρό λόγο. Ίσως είναι μια καλή ιδέα για το μέλλον αυτό. καλό θα ήταν να διαμορφώσουμε με περισσότερα χαρακτηριστικά και περισσότερε περισσότερες λεπτομέρειες αυτή την πρόταση. Αυτά προς το παρόν εμείς είμαστε ανοιχτοί και στην επίτευξη συμβαστικής λύσης και ε, στην έναρξη ε, και συνέχιση του διαλόγου. Εάν δεν θέλει η συγγήτρια να πάρει το λόγο, να δώσει το λόγο στην κυρία Γιατεμάκη. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω το εξής. Οι πωλήσει όπλων στη Φιλανδία είναι ένα θέμα που συζητήθηκε εκτενώς πρόσφατα, διότι μεταξύ άλλων μια μη κυβερνητική οργάνωση δημοσίευσε μια έκθεση η οποία ε, χθες μάλιστα ασκούσε έντονη κριτική ως προς το θέμα αυτό. Βλέπουμε ότι παρακάθηκαν με διάφορους τρόπους οι κανόνες ως προς το εμπόριο όπλων από πλευράς ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο λόγια μπορώ να πω ότι ο έλεγχος των εξαγωγών όπλων δεν, είναι, ε, δεν λειτουργεί με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Δηλαδή, θα πρέπει ε, από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. όπως και ο Πρόεδρος, και εγώ με τη σειρά μου δυστυχώς δεν κατάφερα να τα διαβάσω όλα λεπτομερώς, διότι ε, ήρθε αργά το μεταφρασμένο κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα με δύο λόγια να σχολιάσω τις τροπολογίες που αναφέρονται στην κοινή θέση ως προς το εμπόριο όπλων δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εκεί, σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετήθηκε ψήφισμα ε, πέρυσι. Ωστόσο, με τις τροπολογίες που έχω εγώ υποβάλει, επιθυμώ να πετύχουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ της, μέσα στην έκθεση αυτή. Η κυρία Λόιζιν μας παρουσίασε τη δική της θέση και είναι πολύ έγκυρες οι παρατηρήσεις της. Όμως, εγώ έχω υποκλίνουσα γνώμη ως προς το εδάφιο 27, κυρίες, διότι το ερμηνεύω διαφορετικά. Η κυρία Λοέζη απαιτεί ένα σχέδιο ώστε η παραγωγή στρατιωτικών ε, προϊόντων να μετατραπεί σε παραγωγή προϊόντων για πολιτική, για πολιτική χρήση, για πολιτικούς σκοπούς. Αναφέρεται ότι η επιβίωση του κλάδου είναι πολύ σημαντική στην Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά ε, την δυνατότητα την παραγωγική δυνατότητα στην Ευρώπη, παραγωγή στρατιωτικού υλικού δηλαδή. Και βλέπουμε ότι οι αγορές εξελίσσονται ε, με την κρίση αρνητικά, συρρυκνούνται καλό θα ήταν να συρρυκνωθούν και για άλλους λόγους, όχι μόνο λόγω κρίσης. Για λόγους ειρήνης, επειδή υπάρχει ειρήνη να μην χρειάζεται να, μην χρειάζεται να παράγουμε τόσα πολλά όπλα. Και βλέπουμε ότι όταν ε, δεν τα δίνουμε για τη δική μας άμυνα, τα παρέχουμε στις χώρες τις τρίτες. Όμως θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες ελέγχου και θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες αυτοί οι οποίοι είναι ισχύ αυτή τη στιγμή. Μπορεί η κοινή θέση να μην έχει πάρει τη μορφή οδηγίας ή κανονισμού, παρόλα τα αυτά παραμένει κάτι το δεσμευτικό για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, ε, πιο ανοιχτή στάση. Έχει δίκιο η κυρία Λέζιν και συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει και με τον συνάδελφο Σαν Πέδρο Τέχο προτείνουμε τη συμπλήρωση της κοινή θέσης με έναν δημόσιο κατάλογο ανάλογα με την κατάσταση σε κάθε χώρα μέλος όπου βλέπουμε ότι θα πρέπει να απαριθμούνται οι αρμόδιοι οργανισμοί αλλά και οι χώρες εξαγωγής και να έχουμε και μια αποτίμηση της κατάστασης των αποδεκτριών ε, χωρών, δηλαδή ε, τι συγκρούσεις υπάρχουν εκεί και ούτω καθεξής. Όλα αυτά να συνδέονται με την ε, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έρχονται σε αντίφαση με την πολιτική για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγωγές των όπλων μας θα πρέπει να συνάδουν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική δράση. Όταν γίνεται λόγος για εμπάργο όπλων στη Συρία, ε, βλέπουμε τι θα συμβεί. Είναι κάτι που θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα άλλωστε. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και είπατε εκπρόσωπο, είναι αρμόδια για τη συνοχή μεταξύ ε, της ε, κοινής Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να παρουσιάσω όλες τις τροπολογίες που έχω υποβάλει γραπτός. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, διότι της ανέφερε. Και θέλω να συγχαρώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Εάν προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας και αν ακούσουμε πραγματικά την τεκμηρίωση πίσω από κάθε επιχείρημα, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ε, πολύ καλή έκθεση, η οποία ασχολείται με ένα ζήτημα εξαιρετικά λεπτό και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να συμφωνήσουμε και να πετύχουμε συμβιβαστικές λύσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποφύγουμε κάθε τι που ε, θα ε, πλησίαζε ή θα άπτετο ε, ιδεολογικών ή πολιτικών τοποθετήσεων. Ε, ένα παράδειγμα είναι η τροπολογία 169 169, η οποία δίνει την αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει ή προτείνει να αποφευθεί η παραγωγή όπλων ως γενικότερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την έννοια, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να πω ότι ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το στόχο ως πολίτης το λέω αυτό, διορθώνω, αλλά ως πολιτικός δεν ξέρω αν μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή. Γιατί αν διακόψουμε την ε, παραγωγή όπλων, ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα όπλα αυτά δεν ε, χρησιμοποιούνται μόνο για την επιδίωξη ιδεολογικών στόχων, αλλά και για την επίτευξη της ασφάλειας όπως άλλωστε υπόθηκε και από άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα ικανοποιητικό για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Είναι κάτι που υπάρχει στην Ευρώπη, το γνωρίζουμε, το οποίο άλλωστε το εγγυάται το κοινοτικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι να γίνεται αναφορά ε, στους κανονισμούς και τις ε, διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Δεν θα ήθελα να συνεχιστεί η χρήση του όρου αρνητικός κατάλογος, διότι ε, είναι περιοριστική η ορολογία αυτή για ορισμένες χώρες. Ορισμένες χώρες έτσι φρονούν ότι αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά περιοριστικό. Και είναι σημαντικό να δούμε και τι γίνεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ. καλό θα ήταν να γνωρίζουμε όλοι πόσο λεπτό ζήτημα είναι αυτό που υπάρχει εδώ. Να πετύχουμε συμβιβαστική λύση και να αφήσουμε κατά ιδεολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέρχο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω φιλανδικά. Είχα την ευκαιρία Εν συντομία, να διαβάσω την έκθεση αυτή σε κάποιο βαθμό και πιστεύω ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις είναι πράγματι επικοδομητικές και ελπίζω να είμαστε σε θέση να καταφέρουμε μια συμβιβαστική λύση και μάλιστα γρήγορα και να επιδείξουμε πνεύμα συνεργασίας. Δεν θέλω να εμβαθύνω ε, σε όλες τις λεπτομέρειες των τροπολογιών που έχω υποβάλει. Θα ήθελα να αναφέρω την ε, περιραίουσα αρχή που κρύβεται πίσω από τις τροπολογίες μου. Βασικό στοιχείο είναι η ανάληψη ευθύνης και η διαφάνεια. Ο έλεγχος των εξαγωγών όπλων είναι ουσιώδους σημασίας, είναι απαραίτητος και θα πρέπει να είναι και συνεκτικός, να παρουσιάζει συνέπεια. Ε, επ' αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Οι θέσει εργασία στη στρατιωτική βιομηχανία, στην βιομηχανία των εξοπλισμών είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι θέσει εργασία. Στηρίζουμε λοιπόν ε, αυτό το κλάδο, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτό το στοιχείο της ανάληψης ευθύνης και ελπίζω οι συμβαστικές λύσεις να είναι επικοδομητικές. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν το λόγο, θέλουν να θέσουν ερωτήσεις ή κάτι άλλο. Όχι, η κυρία Λέζη να θέλει να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξαναμπώ σε όλα όσα είπα. Να καταστήσω σαφές ότι πρόκειται για την μεταγραφή της κοινή θέσης, την εφαρμογή της. Κάποιοι συνάδελφοι στην τελευταία συζήτηση είπαν ότι θέλουν να την τροποποιήσουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η ε, άποψη των περισσότερων. Θέλουμε να εφαρμόσουμε βεβαίως την κοινή θέση με βάση κάποια κριτήρια βεβαίως για τον έλεγχο των εξαγωγών εξοπλισμών. Βεβαίως υπάρχουν ε, αντιθέσεις συμφερόντων, άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης να ε, εξεύρουμε συμβασμούς και να μπορέσουμε ε, να εφαρμόσουμε στο μέλλον λοιπόν την κοινή θέση. Έλαβα κάποιες συμβολές και από τις εκκλησίες. Ίσως λοιπόν να διευκολύνει κάποιους να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν κάποιες θέσεις. Κάποιες προτάσεις των εκκλησιών ήταν ε, πιο συνεπείς και πιο ριζοσπαστικές από τις αρχικές μου θέσεις και τις έλαβα υπόψη γιατί καταδεικνύουν και την ηθική διάσταση της έκθεσης, την ηθική διάσταση των, αποφάσε των αποφάσεων που θα πάρουμε για το α ή β θέμα. Ναι μεν κατέστησα σαφές ότι η πολιτική μας κατεύθυνση είναι υπέρ μιας μετατρο... μετατροπής των ε, βιομηχανιών όπλων, αλλά σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να θέσουμε κανόνες για την εξαγωγή εξοπλισμών. Αυτό και μόνο είναι το καθήκον μας τώρα. Ευχαριστώ. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Όπως βλέπετε, όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ήταν από τη Φιλανδία και την Πολωνία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο χώρες αυτές είναι και οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς όπλων. Τώρα, ε, να σας πληροφορήσω για το εξής. Ε, δεύτερη ανάγνωση και υιοθέτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 27 Απριλίου και συζήτηση στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα. Επομένως μένει ακόμα χρόνος για συνομιλίες και για την επίτευξη συμβιβασμών. Πάμε τώρα στη δεύτερη μας έκθεση το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Γιαννάκου για τις ε, στρατιωτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σήμερα έχουμε το τελικό κείμενο της έκθεσης. Ε, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία για την πολύτιμη βοήθειά της στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής ε, και τη συμβολή της νομίζω σε μια καλή προσπάθεια. Ε, θέλω να σας πω πριν να, γίνει η έκθεση ότι είχα μια συνάντηση ε, με τον στρατηγό Βανός του στρατιωτικού επιτελείου καθώς και επαφές με το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το European Defense Agency. Ε, θα επαναλάβω ότι η έκθεση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη συνολική προσέγγιση της Ένωσης ούτε προσπαθεί να υπερτονίσει μόνο κάποιες επιμέρους διαστάσεις έναντι άλλων. Ε, αυτή την επισήμανση την έκανα και στην πρώτη συζήτηση που είχαμε πριν λίγες μέρες και θα πρέπει να γίνει κατανοητή ώστε να μην εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις για τη φύση της εξωτερικής δράσης ε, αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση στο τμήμα της ανάπτυξης καθαρά στρατιωτικών ικανοτήτων σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που είχε αποκτήσει πριν από δέκα περίπου χρόνια. Σαφέστατα η προσπάθεια αυτή λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεχών περικοπών στους αμυντικούς προϋπολογισμούς γίνεται πιο δύσκολη ακόμα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό του αμυντικού σχεδιασμού. Οι συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη λύση στα προβλήματα που επιβάλλει το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που χρειάζεται η Ένωση για να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις της στη διεθνή ασφάλεια και στη διαχείριση κρίσεων. Αυτό που επιδιώκεται είναι να ενδυναμωθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η έκθεση κινείται στους εξής άξονες, γενικές παρατηρήσεις, στις δομές σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατιωτικών επιχειρήσεων, τις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, στις μόνιμες πολυεθνικές δομές των κρατών μελών, στην ανάπτυξη δομών και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών αδυναμιών της Ένωσης, στην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και τις ασκήσεις, στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και στην αναβάθμιση της ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι γεγονός ότι η έλλειψη ενός επιχειρησιακού στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων δυσχεραίνει την ετοιμότητα της Ένωσης να αντιδράσει αποτελεσματικά και έγκαιρα στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Η ενεργοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων για τον συντονισμό των αποστολών στο κέρας της Αφρικής αποτελεί ασφαλώς το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Εν τούτης το κέντρο αυτό δεν είναι ούτε μόνιμο, ούτε αποτελεί κεντρικό σημείο σχεδιασμού και διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η στελέχωσή του παραμένει ακόμα ανεπαρκής. Η δημιουργία ενός μόνιμου επιχειρησιακού στρατηγίου θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής κουλτούρας και θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μακροπρόθεσμα θα επιφέρει λιγότερες δαπάνες και θα διευκολύνει τον πολιτικό έλεγχο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να υποτιμάται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για αυτούς τους λόγους η ίδρυση ενός επιχειρησιακού στρατηγίου είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Οι δυνάμεις ταχείας αντίδρασης. Όλοι μας αναγνωρίζουμε τη συμβολή των ευρωπαϊκών δυνάμεων ταχείας αντίδρασης, των battle groups, στο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών, στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και στην πρόθεση της πολυεθνικής συνεργασίας. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι ως σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα από τα EU Battle Groups, αν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δύναμη πρώτης εισόδου σε αρκετές περιπτώσεις. Αποδεικνύονται λοιπόν οι δομικές αδυναμίες στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών. Είναι προφανές ότι το τωρινό πλαίσιο δεν λειτουργεί Πρέπει να αναζητήσουμε όλους τους πιθανούς τρόπους για την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης και κυρίως να ενθαρρύνουμε την πολιτική βούληση των κρατών μελών για να το χρησιμοποιήσουν. Κατά την άποψή μου δύο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Το ένα είναι η χρηματοδότηση και το άλλο είναι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ενεργοποίησή τους. Ακόμη και ο αναθεωρημένος μηχανισμός Ατένα δεν λαμβάνει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των EU Battle Groups και πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό των κοινών δαπανών διασφαλίζοντας επομένως το δικαιότερο επιμερισμό της επιβάρυνσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ένα dedicated fund για τη χρηματοδότηση των battle groups θα μπορούσε να είναι μια λύση. Ακόμα πιστεύω ότι τα κόστη που δεν συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτές καθ' αυτές, όσα δηλαδή αφορούν την προετοιμασία και τη διατήρηση των battle groups θα μπορούσαν να καλυφθούν απευθείας από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διότι αυτό το τμήμα δεν το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Ε, όσο αφορά στη λήψη αποφάσεων, είναι γεγονός ότι μας χρειάζεται πιο μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους απόδοσης κάποιων περιορισμένων εξουσιών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην ύπατη εκπρόσωπο για την ενεργοποίηση των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον βέβαια εκπληρούνται κάποιες σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις. Στο κομμάτι ανάπτυξης δομών και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των σημερινών αδυναμιών μας χρειάζεται μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση σε τομείς όπως στρατηγικές αερομεταφορές, ελικόπτερα, ιατρική βοήθεια κτλ. Άρα τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθήσουν συστηματικές αναθεωρήσεις στους τομείς ασφάλειας και άμυνας με βάση εναρμονισμένα κριτήρια. Σε αυτό το πεδίο η συνεκμετάλλευση και ο επιμερισμός ικανοτήτων, το pooling and sharing, δεν αποτελεί επιλογή, αλλά επίγουσα αναγκαιότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντική θα είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εναρμονίσουν τους αμυντικούς σχεδιασμούς, σύμφωνα με το Capability Development Plan της ε, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας. Υπάρχουν ήδη σημαντικά παραδείγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και οφείλουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Η κοινή ιδιοκτησία, παραδείγματο χάρη κάποιων ακριβών ικανοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για μη στρατιωτικέ χρήσει, είναι μια επιλογή που πρέπει να την προωθήσουμε. Δυστυχώς ως σήμερα δεν υπάρχει σαφής δέσμευση από πλευρά κρατών μελών για την ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων. Και γι' αυτό το λόγο η ύπατη εκπρόσωπος πρέπει να παρουσιάσει νέες σαφείς προτάσεις. Παράλληλα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια παροχής του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων και να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη εξάρτηση από τις μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες οι οποίες είναι και ακριβές από τις μη ευρωπαϊκές δηλαδή πηγές εξοπλισμού εδώ έρχεται το θέμα της προστασίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνογνωσίας, η οποία α, χρησιμοποίηση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη αυτού του στόχου. Πέρα βέβαια από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη είτε διμερώς είτε μέσω συμμετοχών σε πολυεθνικούς σχηματισμούς Αυτές οι δράσεις πρέπει να συντονιστούν υπό την αιγίδα ενός συνολικού σχεδιασμού και όχι να περιοριστούν. Στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπαρχουσών πρωτοβουλειών και σε αυτό το σημείο πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί με την EU Military Committee αλλά και η αξιοποίηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Επιπλέον πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση της εξειδίκευσης και των κοινών ασκήσεων της Ευρώπης. Ο ρόλος του European Security and Defence College είναι σημαντικός, όπως επίσης και κάποιων άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, όπως το πρόγραμμα Έρασμους. Δεν έχει αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτή η προσπάθεια. Τώρα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ θα πρέπει να επισημάνω τη φιλοδοξία της Ένωσης για την σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινή αμυντικής πολιτικής. Σέβεται τις υπάρχουσες συμμαχίες, ιδίως στο ΝΑΤΟ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε τις προσπάθειες προώθησης μιας στρατηγικής αυτονομίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων από την Ένωση θα ωφελήσει και το ίδιο το ΝΑΤΟ πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαλειτουργικότητα και τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν και αυτό θα μας βοηθήσει και στην υπόθεση της περικοπής των προϋπολογισμών. Το τελευταίο κομμάτι της έκθεσης αναφέρεται στις μελλοντικέ προοπτικές και ιδιαίτερα στο θέμα της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και να κάνουν ένα βήμα μπροστά στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Επί του παρόντος, ο ορισμός της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας μπορεί να φαίνεται κάπως δύσκολος, λόγω του ότι υπάρχουν διαφωνίες ακόμα σε επίπεδο Συμβουλίου. Ωστόσο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τίποτα δεν μας εμποδίζει να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η έκθεση δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία είναι και φιλόδοξα αλλά και ρεαλιστικά. Στοχεύουν στην ενισχυμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και στην ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της διαρθρωμένης συνεργασίας. Σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταλήξω και να ζητήσω και την άποψη των συναδέλφων για το θέμα της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιους σκιώδε εισηγητέ εισηγητές στην αίθουσα. Κύριε Πάσκο, έχετε το λόγο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι είναι λίγα τα μέλη εδώ, η σημασία του θέματος δεν μπορεί ούτε να αγνοηθεί ούτε να παραμεληθεί. Και νομίζω ότι γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε στο εξή σημείο. Αν συνεχίσουμε στο δρόμο που έχουμε ήδη πάρει, πολύ γρήγορα θα φτάσουμε στο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή δυστυχώς. Και είναι δικό μας καθήκον να το επισημάνουμε αυτό και να καταδείξουμε τη δική μας άποψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ότι δηλαδή χρειάζεται να αναχαιτιστεί αυτή η τάση και να επανέλθουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη χάνει όλο και περισσότερο έδαφος. Εκχωρούμε υλική δύναμη σε άλλους, πουλώντας πλατφόρμες, ε, οπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μη επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη και έτσι χάνοντας το τεχνολογικό πλεονέκτημα, μειώντας πλέον σε θέση παραγωγής τεχνολογίας εχμής, και παρόλο που θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη διεθνή αρένα, ε, χάνουμε έδαφος και είναι περίεργο να λέμε ότι η φιλοδοξία μας είναι να αποκτήσουμε στένος περισσότερο, ενώ χάνουμε όλο και περισσότερο έδαφος. Δεν ξέρω. Ε, στην ουσία αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να ε, πούμε ως εδώ. Και η έκθεση αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει. Ο πρόεδρος Μπαρόζο για πρώτη φορά στην ε, δήλωση που έκανε στην αρχή της χρονιάς για την κατάσταση της Ένωσης ε, είχε μία παράγραφο για το θέμα αυτό αναφερόμενο στα σημεία που έχουμε ήδη συζητήσει, αν καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις, οι οποίες μπορεί εν μέρη να φαίνονται επαναστατικές και μη αποδεκτές για τον τρόπο με τον οποίο αλληλοπεδρούν τα κράτη στο Συμβούλιο, τότε είναι καθήκον μας να το πούμε. Να ζητήσουμε από τους άλλους να τους κρίνουν και να τους καλέσουν να προβληματιστούν. Ίσως κάποιες χώρες θεωρήσουν ότι δεν είναι τόσο μη αποδεκτά ή απαράδεκτα μέσα από τα πράγματα και θα μπορούσε να υπάρξει μια, ε, κάποια πρόοδος εκεί. Και πέρα από το Συμβούλιο υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει την αλλαγή στις συνθήκες. Γιατί να αφήσουμε να πάει χαμένη μια τέτοια ευκαιρία και να περιμένουμε να ανακύψει μια άλλη ευκαιρία την οποία ε, δεν γνωρίζουμε η οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα δημιουργηθεί και δεν ξέρουμε και τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει τέτοιου είδους εξελίξεις. Ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να στοχεύει στην ενθάρρυνση της πολιτικής βούλησης, γιατί το βασικό ερώτημα δεν είναι τόσο τεχνικό το βασικό ζήτημα, βεβαίως μπορεί να είναι οικονομικό, αλλά ταυτοχρόνως η πολιτική βούληση έχει την ίδια, αν όχι και μεγαλύτερη σημασία. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο αυτές τις ε, ομάδες και μονάδες ταχείας αντίδρασης. οι οποίες όταν τις παρουσιάζουμε φαίνονται τέλειες, αλλά όταν ε, έρχεται η ώρα της αξιοποίησής τους, κανείς δεν θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω αυτή την ιδέα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προσφεύγει σε ένα τέτοιο είδους μέσο όταν το χρειάζεται, μαζί και με το Startup Fund, κάτι το οποίο το τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται αυτές οι δράσεις και επιχειρήσεις, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Ακόμα και αν ε, το κάνουμε μόνο για να στερήσουμε από τους άλλους τη δυνατότητα να προβάλλουν εμπόδια οχυρωνόμενοι πίσω από την υποτισέμενη τεχνική δυσχέρεια ενώ ουσιαστικά τους λείπει ε, πολιτική βούληση. Τώρα, έχουμε αυτό το κέντρο αποθήκευσης για το ε, Capability Development Plan και για, το, για την κοινή ε, πολιτική ασφάλειας. Έχουμε το EuroCorp που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί στο Αφγανιστάν. Έχουμε δηλαδή ένα πυρήνα και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να ε, επιταχύνουμε, να δώσουμε όθηση στα πράγματα, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος. Κυρία Νικολάη. θεωρούμε ότι η έκθεση είναι μια πολύ καλή αρχή. Πρέπει να επεκτείνουμε την έκθεση αυτή. Πρέπει να την επεκτείνουμε και μπορούμε. Και πρέπει να έχει βασικές ρωμαλές και σαφείς ιδέες. Για μένα το κύριο θέμα είναι το μέλλον της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, όχι απλώς ε, η κατάσταση και οι προοπτικές. Αυτή είναι η στόχη της κοινή μα πολιτικής. Της κοινής μας πολιτικής. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι και αν θέλουμε να ακουστούμε, αν θέλουμε να περάσουν οι ιδέες μας, πρέπει να υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί στις συνθήκες. Έχουμε πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφε, με τις συνθήκες. Αν δούμε το άρθρο 41 μόνιμη δομή συνεργασία αναφέρεται εκεί συνέχεια. Αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν είναι πολλές οι χώρες που θέλουν και είναι σε θέση να υπάρξει αυτή η διαρθρωμένη συνεργασία. Πολλά κράτη-μέλη αποφεύγουν να εργαστούν στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που επιτρέπεται από τις συνθήκες. Ίσως γιατί όλοι έχουμε ακούσει ότι μπορεί να τροποποιηθεί η συνθήκη. Ίσως λοιπόν να πρέπει να αρχίσουμε την προσπάθεια για πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις στον τομέα της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας άμυνας. Είναι μια καλή αρχή, εάν καταλήξουμε ότι έχουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της κοινή πολιτικής ασφάλειας άμυνας, να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την ε, μάχη. Γιατί υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά ε, καμία δεν πηγαίνει όσο μακριά πρέπει. Η έκθεση δεν έχει προήμιο, αλλά θα έπρεπε να εξηγήσουμε στο κείμενο ότι τα θέματα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Πρέπει επίσης να εξηγήσουμε σαφώς γιατί θέλουμε πιο μόνιμη δομή και να αναλογιστούμε πώς θα αξιοποιήσουμε πολυμερός εάν δεν συμφωνούν όλοι αυτές τις ε, δομές. Θέλουμε ένα μηχανισμό για να μπορεί κανείς να εξαιρεθεί, opt-out, για παράδειγμα για τα, μία ζωτικά, για τα μη ζωτικά στοιχεία μιας αποστολής ή να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εκπεριτροπής. Συνέχεια όμως πρέπει να συνδυάζουμε και να χρησιμοποιούμε από κοινού pool and share τις ικανότητές μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εργαστούμε στον τομέα της άμυνας. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή μας την πείρα και για τη διαχείριση θεομηνιών. Πρέπει βεβαίως ε, να συζητήσουμε το θέμα αυτό για να καταλήξουμε σε σαφές όραμα για το ποιος θα συντονίζει τα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο και εάν, ε, διατηρήσουμε την, ε, εάν θα διατηρήσουμε την υπάρχουσα δομή ή όχι, γιατί πρέπει να την αποτιμήσουμε σε αυτή τη φάση, την παρούσα δομή και ίσως να προτείνουμε κάτι πιο θαραλέο. Τέλος, τονίζω, ότι αναφερόμεθα συνέχεια στην οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της ε, στον τομέα της άμυνας και συνέχεια εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μία αντίδραση μέσω της έκθεσης για να απαντήσουμε στα εξής τρία θέματα. Να χρησιμοποιούμε όλα όσα έχουμε εγώ θα έλεγα ότι δεν το κάνουμε πάντα. Δεύτερον, πρέπει να επενδύσουμε ως Ένωση σε όλα τα μέσα που έχουν διάθεσή μας. Και το τελευταίο, θέλουμε ένα κοινό πόρο ως στρατιωτικό δυναμικό. Έτσι πιστεύω εγώ και νομίζω ότι έτσι πιστεύετε κι εσείς. Καλή αρχή λοιπόν η έκθεση αυτή και θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες και από μένα και από την ομάδα μου Άλντε. Πρόεδρος, η κυρία Λόζιν. Συμφωνώ σε αυτά που είπε ο κύριος Πάσκο. Συγκεκριμένα είπε ότι υπολείπεται συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και μειώνεται η επιρροή της και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να το πούμε και εδώ και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί ε, ναι μπορεί για ορισμένες, ε, σε ορισμένες πλευρές να ισχύει αυτό, αλλά δεν ισχύει για άλλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Εγώ νομίζω ότι δεν άξιζε να το πάρει. Πιστεύω ότι πρέπει να εργαστεί περαιτέρω σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να βαδίσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε αξιοπιστία. Αυτός θα ήταν ο δρόμος για να γίνουμε πιο πιστευτοί. Κυρία Γιαννάκου. Η έκθεση είναι φιλόδοξη, θεωρείται φιλόδοξη. Είναι όντως πολύ φιλόδοξη. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα σημεία, αλλά η απόλυτη υποχρέωση σε σχέση με την ρήτρα αλληλεγγύης είναι να αντιμετωπίζουμε από κοινού τις απειλές σε μια συγκυρία όπου παγκόσμια συζητείται η ηθική χρήση αυτών των όπλων. Συνεργασία αλλά και αυτονομία από τον ΝΑΤΟ και το, το σύστημα Γαλιλαίος για στρατιωτικούς στόχους. Οποτεδήποτε είχα ε, ισχυριστεί κάτι στο παρελθόν μου είπαν όχι κυρία Λόζινγκ δεν είναι αλήθεια. Ε, μόνο για μη στρατιωτικού στόχους χρησιμοποιείται το Γαλιλαίο. Να λοιπόν που η έκθεση το αναφέρει τώρα σαφώς. Είναι σαφές προς ποια κατεύθυνση εγώ και η ομάδα μου πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Η έκθεση, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι κατά τη γνώμη ένας κατάλογος όλων των στόχων που θα έπρεπε να επιτευχθούν για να παίξει ουσιαστικά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση στον τομέα αυτό. Οπότε πρέπει να γίνει μια μεγάλη ζήτηση για αυτό βέβαια, αλλά δεν έχουμε καμία διαφωνία επί τη ουσία, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί την ειρήνη και είμαι βαθιά πεισμένη ότι μπορούμε μέσω στρατιωτικής συνεργασίας να επιτύχουμε αυτό. Θα πρέπει όταν επεμβαίνουμε σε ε, διενέξεις να το κάνουμε για να προωθήσουμε την ειρήνη. Και εδώ στη ΣΕΝΤΕ και στην ΑΦΕΤ πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να γίνεται πριν ξεκινάει μια στρατιωτική αποστολή μια αποτίμηση της κατάστασης. Πρέπει να το ζητήσουμε σαφέστατα. Διότι, κατά τη γνώμη μου, καμία από τις στρατιωτικές μας παρεμβάσεις δεν βελτίωσε την κατάσταση του πληθυσμού και δεν κατάφερε να σταματήσει μια στρατιωτική διένεξη. Τώρα, για τις κρίσεις. Πολύ συχνά γίνεται η σύνδεση οικονομικής κρίσης και ε, των απαιτήσεων που θέτει η έκθεση. Εγώ νομίζω ότι είναι κοινικό στην ε, παρούσα συγκυρία που υπάρχει τόση πολιτική λιτότητας που γίνονται τόσες περικοπές που απειλούν την ίδια την επιβίωση των πληθυσμών μας, να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα εμείς θέλουμε να ε, κάνει η Ένωση, την ανθρωπιστική της αποστολή. Και για τη δημοκρατία πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο δεν ελέγχει στην ουσία τις ε, στρατιωτικές παρεμβάσεις και τον ε, προϋπολογισμό άμυνας. Γι' αυτό πρέπει να το καθορίσουμε, να το ε, τονίσουμε αυτό. Χαίρομαι λοιπόν που όπως και εσείς είπατε ότι ακόμη στα ευρωπαϊκά κράτη δεν υπάρχει πλειοψηφία για τέτοιες πολιτικές, ίσως για άλλους λόγους από αυτούς που ανέφερα εγώ. Αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι που όντως ούτως έχει η κατάσταση. Δεν θα σας εκπλήσει ότι απορρίπτουμε πλήρως αυτή την έκθεση και θα υποβάλουμε εναλλακτική ε, έκθεση μειοψηφίες για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γνωριζόμαστε πολύ καλά, δεν μας προκαλεί εντύπωση το συμπέρασμά σας. Ο κύριος Πάσκου επίσης θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι εμείς ουσιαστικά είμαστε υπεύθυνοι, κινητοποιούμε, δίνουμε λόγους για να αυξηθεί ο προπολογισμό. Μάλλον εμείς ουσιαστικά, με συγχωρείτε, μέσω της κρίσης δικαιολογούμε τη μείωση του προπολογισμού. Είναι όμω καλύτερα τα πράγματα έχοντα μειώσει του αμυντικού προπολογισμού μέσω τη κρίση. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά τα οποία περικόψαμε από του αμυντικού προπολογισμού, έτσι ώστε εγώ να αισθάνομαι ότι δεν με πειράζει τόσο πολύ τελικά η οικονομική κρίση. Ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα έχουμε δηλαδή. Λέμε ότι δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε αύξηση του προπολογισμού εξαιτία τη κρίση, αλλά παράλληλα αυτό που βλέπουμε είναι ότι μειώνουμε τον αμυντικό προπολογισμό και δεν, δεν αποφελούμαστε από τίποτα. Δεν ζούμε καλύτερα στο τέλο. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι το επιχείρημα μπορεί να παρουσιαστεί και αντίστροφα στην περίπτωση αυτή. Αντίθετα δηλαδή από αυτό το οποίο γενικότερα λέγεται ότι ε, η οικονομική κρίση ε, δεν μας επιτρέψει καμία περίπτωση να αυξήσουμε τους αμυντικούς προπολογισμούς. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Κύριε Γεννάκου, θέλετε να πάρετε το λόγο για τελευταίες παρατηρήσεις. Ε, ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους <clears throat> για τις παρατηρήσεις τους ε, και βέβαια ασφαλώς ε, εν ώψη του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ε, η έκθεση είναι φιλόδοξη αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια πραγματικότητα δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθήλωση ε, ε, των φιλοδοξιών που είχαν αναπτυχθεί πριν από 10 χρόνια και όσο αφορά στην χρηματοδότηση υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί η περικοπή των προπολογισμών με τις συνέργειες και τις σωστές συνεργασίες. Και αυτό είναι που επιδιώκουμε. Δηλαδή έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε οι οποίες έχουν ένα χι αποτέλεσμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αποτέλεσμα πολύ κατώτερο από αυτό ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν συνέργειες. Δεν σας λέω να γίνουμε ε, Ηνωμένε Πολιτείες πρώτα για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Μπορούμε όμως ε, στο στρατιωτικό τομέα συνδυασμένο με τον ε, πολιτικό τομέα, δηλαδή με τα ζητήματα πολιτικής άμυνας, με τη συμμετοχή της Europol όπως ελέγχθη πριν κτλ. μπορούμε να επιτύχουμε κάλλιστα ε, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επομένως δεν είναι μια οριζόντια υπόθεση έχουμε πολλά χρήματα όλα καλά και έχουμε λιγότερα και δυστυχώς και όταν είχαμε περισσότερα χρήματα δεν πήγαιναν καλά τίποτα. Άρα το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει τις προτάσεις του και νομίζουμε ότι αυτές δεν είναι μονολογικές αλλά προέρχονται και από την εμπειρία των στελεχών. Τα στελέχη που εγώ συνάντησα από τις στρατιωτικές δομές μου είπαν ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα και πιο αποτελεσματικά με κάποιες κινήσεις και αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν αυτά πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι εκεί στοχεύει η έκθεση. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 11η Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 16 Μαΐου. Έγκριση στην συνεδρίαση της ΑΦΕΤ στις 30 Μαΐου και προβλέπεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου η έκθεση αυτή. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις ή άλλα σημεία στη μερίσια διάταξη, λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.